Uh, uh, Φίλοι, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο τμήμα της ε, ψηφοφορίας της εκθέσης ε, του Ζωαβρέρα για τα Ταμεία Συνοχής ε, και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά το διάλειμμα μας λοιπόν, η πρώτη ψηφοφορία θα είναι δύο τροπολογίες, η 235 και η 236, 235 και 236. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται.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 άδικο αυτό που λέτε, λέει ο Πρόεδρος, γιατί ήταν σαφές ότι απορρίφθηκε. Μάλιστα. Δύο τροπολογίες λοιπόν και πάλι. Η 235 και η 236. Ψηφίζουμε. Έναξη ψηφορίας. Πέρας τώρα. Εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα. Εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα και εγκρίνεται. Μα τι κάνετε, λέει ο πρόεδρο. Φίλοι μου. Amendment 284. Η 284, δεύτερο τμήμα. 284, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Μια και δεν συμφωνούμε εδώ με τον Κλάους. Πέρας. Απορρίπτεται και δίκιο έχετε. Η 284 τρίτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδια η πλειοψηφία. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο παρακαλώ για την 239. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κι αυτή. 246 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 287 τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 287 τρίτο τμήμα. 287 τρίτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 287 τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος. Για την 252. Πέρας ψηφοφορίας. 287. Απορρίφθηκε η προηγούμενη. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. ψηφίσετε λίγο ανάποδα σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 286 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης. 250 υπέρ. Κατά. απορχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 251. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. 287. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 287. Έκτο κομμάτι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 288. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 266. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 288 τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 289. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 289. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 290 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος 269. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρασε. Απορρίπτεται. 275 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 278 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 291. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται επίσης. 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 291 τρίτο τμήμα υπέρ κατά Έλαχος για την 291 συμβαστική Κομμάτι τρίτο το τμήμα πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 71. Και πέρας. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 από το τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 75. Πέρας. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Εκ νέου έλεγχος, παρακαλώ. Για την 76 έλεγχο. Και πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται επίση, 77 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Απόχε Εγκρίνεται. Η 5D υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για τροπολογία 80. πέραση ψηφορίας. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται 85 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ή την 87 84 πέρα λέει ο πρόεδρος πέρα στις ψηφορίες και απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά Απόχες εγκρίνεται 11 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται 87 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται 88 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 89 πέρας απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 δι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 94 πέρας απορρίπτεται 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται 97 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται 98 υπέρ. Κατά Έλεγχος για την 98. πέρα Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 102. Πέρασε. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 17. Θέλετε έλεγχο. 17 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Ζητείτε έλεγχο. Άντε για να ξυπνήσουμε, λέει ο πρόεδρος. Για την 104 παρακαλώ. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται 106 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται 107 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται 19 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται 20 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 58 η 58 τη θυμάστε δεν τη ξεχάσατε, πριν από λίγες ώρες την είχαμε υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε αυτή την ιδιαίτερη τροπολογία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Όπως έχουν εγκριθεί οι τροπολογίες, με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚΑ. Μάλιστα. Απορρίπτεται. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι σαφές. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ε, ο εισηγητής είναι ο κύριος Φέντερλη. Ε, λειτουργία του ονόματος τομέα ανώτατου επίπεδου ΥΓΙΟΥ. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ο Πολ Ρούμπιχ ε, δεν είναι μαζί μας, γι' αυτό κανείς δεν ζητά ονομαστική. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία στο σχέδιο όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική. Okay, I close the vote. Πέρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη υποστήριξη. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αγαπητοί φίλοι. Αγαπητοί φίλοι. Έχουμε ε, τη δεύτερη ψηφοφορία πάλι με ονομαστική κλίση. Κύριε Φέντερλε, ακόμα πιο σημαντική αυτή η ψηφοφορία γιατί πρόκειται για τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Ψηφίζουμε. Πέρας. Συγχαρητήρια, κύριε Φέντερλε. Τώρα πρέπει να είσαστε απόλυτα ικανοποιημένος. Λοιπόν, Λοιπόν, κανονισμός για τη δίκαιη μεταχείριση και διαφάνεια για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. <clears throat> δηλαδή πλατφόρμες στην ουσία. Η κυρία Ναζαμπόρσκα είναι η εισηγήτρια ο Πολ Ρούμπιχ δεν είναι εδώ. Προχωράμε λοιπόν ακάθεκτη. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 9, υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 10, υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 11, υπέρ κατά αποχές Δεχτεί Κανένας βλέπω δεν ψηφίζει. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3.47. 3.47. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 3.47. 3.47. Ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.48 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε και την 3.48. Ας έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη, την στη χαρά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.53 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά ας ελέγξουμε λοιπόν την 50 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 55-56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 62 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 62, έλεγχος. Μπορείτε ακόμα να ψηφίσετε. Ψηφίζουν 54, όχι 67. Πέρας. Απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 131 υπέρ, κατά, αποχές αποδεκτή, 112 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 129 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και τώρα τελική ψηφοφορία με ονομαστική τελική ψηφοφορία για σήμερα. Πέρας. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα συνεχίζουμε κανονικά με την Επιτροπή, με τις εργασίες της Επιτροπής. Μπορείτε να παραμείνετε αν θέλετε. Η κυρία Νίμπλερ είναι παραούσα. Ωραία. Συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας, αν και αν μειώθηκε ο αριθμός μας. Θα σας πρότεινα λοιπόν να αρχίσουμε με τα πρακτικά από την κυρία Νίμπλερ για το θέμα της ε, ρομποτικής ε, και της ασφάλειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι, να σας στηρίσω λίγο ενήμερους με τη, σε σχέση με το τι έχει γίνει. Ε, κάναμε τρεις ε, τρεμερείς διαλόγους για την ασφάλεια και προχωρήσαμε, προχωρήσαμε μια χαρά. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα λάβει χώρα ο τέταρτος τρεμερείς διάλογος, ο οποίος θα διαρκέσει μόλις μια ώρα. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα πράγματα, αλλά προληπτικά προβλέψαμε και μία συνεδρίαση το Δεκέμβριο, μπας και χρειαστεί. Έχουμε δύο βασικά τμήματα. Καταρχάς έχουμε τα καθήκοντα και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ΕΝΙΖΑ για την κυβερνοασφάλεια. Κάναμε πολλές πρόοδους εδώ σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της ΕΝΙΖΑ, τη συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τα ρυθμίσαμε όλα αυτά. Στο δεύτερο βασικό τμήμα της πρότασης έχουμε το θέμα της πιστοποίησης. Εδώ είμαστε λίγο ε, σε πιο εκρεμή θέση υπάρχουν και διαφορές σε σχέση με την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, το θέμα της συνεργασίας, της κατανομής των αρμοδιοτήτων, θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να καταφέρουμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Έχουμε υποβάλει τι προτάσει μα. Το κατά πόσο βέβαια θα το πετύχουμε, αυτό εξαρτάται και από τα κρατημέλη και από την προθυμία που θα δείξουν και αυτά να απαντήσουν στι ε, αξιώσει μα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και ελπίζω να καταφέρουμε να το κλείσουμε το θέμα αυτό υπό Αυστριακή Προεδρία. Αυτό είναι Άλλωστε, ο στόχο όλη ε, τη αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, αυτό ασφαλώ δεν είναι εξαρτάται μόνο από εμά, εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Για να ολοκληρώσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα, θέλουμε, ότι, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ενίζα να καταστεί μια αυτόνομη, δυναμική ε, οργάνωση, ε, αυτόνομος ε, Δυναμικό Οργανισμό και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πετύχουμε καλέ λέξει. Να ευχαριστήσω και όλους τους κοιότητες συζητητές, ε, να τον τονίσω αυτό και ο κύριο Τέλτσκα είναι εδώ. Δεν βλέπω του άλλου συναδέλφου. Νομίζω ότι ω αντιπροσωπεία ήμασταν πολύ δυναμικοί, ενωμένοι, παρουσιάσαμε καλά επιχειρήματα και νομίζω ότι πραγματικά υποστηρίξαμε τη θέση μας και αν έχετε ρωτήσει φυσικά να σας τις απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα ήθελα οι σκιώδεις να ε, λάβουν το λόγο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ο, ο κύριος ε, Τέλισκα, στην ουσία το μπαλάκι είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Εν πάση περιπτώσει ε, όλες οι διαπραγματεύσεις κινήθηκαν σωστά και θα δούμε κατά πόσο το Συμβούλιο θα, έχει, θα μας αφήσει περιθώριο ελιγμών. Εν πάση περιπτώσει υποστηρίζω την εισηγήτρια σε αυτή τη την προσπάθεια. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, δεν νομίζω ότι είναι η περίπτωση. Ε, τελειώνουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, πιστεύοντας ε, ε, αίσιου πέρας. Ashley Fox ε, στη συνέχεια θα δούμε το επόμενο σημείο σε σχέση με την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική ε, αποτελούν ένα κρίσιμο ζήτημα ε, για τις χώρες μας τα επερχόμενα χρόνια και είναι ένα θέμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει εγκαίρως. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι αυτή η έκθεση προτάθηκε για πρώτη φορά από τη Γραμματεία το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Και το Κοινοβούλιο μετά δαπάνησε έξι μήνες λογομαχώντας για το ποιες επιτροπές, ποια η επιτροπή είναι η καθήλυν αρμόδια και ούτω καθεξής. Άρα ανατέθηκε τον Οκτώβριο η έκθεση και έτσι οι επτά εμπλεκόμενες, εμπλεκόμενες επιτροπές δεν μπορούν να παράσχουν στοιχεία που να έχουν ε, αξία. Η, ε, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, το Bundestag και η Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αποφανθεί Μιλάμε για 238 σελίδες ως προς τη ε, Βουλή των Λόρδων. Η δική μου έκθεση είναι ταπεινή, αφορά γύρω στις έξι σελίδες. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να δούμε πώς το Κοινοβούλιο θα φτάσει σε ένα συνεκτικό και αξιόλογο έγγραφο, γιατί υπάρχουν ε, δύο άλλε επιτροπέ με αποκλειστική αρμοδιότητα επί του θέματος. Θα έχουμε και άλλε γνωμοδοτήσει. Θα συναντηθώ με τον κύριο Μπούζεκ αργότερα σήμερα και ελπίζω να επεκτείνουμε κάπως το χρονοδιάγραμμα, διότι αυτή τη στιγμή Έχουμε προθεσμία την 6η Δεκεμβρίου για τις τροπολογίες και ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 7 Ιανουαρίου, δηλαδή μία μέρα μετά την επιστροφή μας. Ε, δεν είναι τρόπος λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αν θέλουμε να μας παίρνουν σοβαρά υπόψη πώς επιτρέψαμε στους εαυτούς μας να χάσουμε έξι από τους εννέα μήνες λογομαχώντας για το ποια επιτροπή θα αναλάβει τι. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Και ένα κοινοβούλιο που συμπεριφέρεται έτσι δεν αξίζει να εισακούεται. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς που εργαστήκαμε σε αυτή την έκθεση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να φτάσουμε σε κάτι ουσιώδες. Έχετε το ε, σχέδιο γνωμοδότησης, ένα μικρό έγγραφο, δεν λέει και πολλά, αλλά αυτό γιατί ε, δεν υπήρχαν περιθώρια. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάτι το ουσιώδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία πραγματιστική ε, προσέγγιση ως προς την τεχνητή νοημοσύνη και οι έρευνες που διενεργούνται γίνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις γιατί φυσικά έχουν κέρδος σε σχέση με το κεφάλαιο που επενδύουν και έτσι πρέπει να έχουν τα πράγματα. Και πολλές εθνικές κυβερνήσεις θα θέλουν να ταχθούν επικεφαλής αυτής της τεχνολογίας στη δική τους χώρα, κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς δεν θα υπάρχει ειδική ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κανένα κράτος μέλος δεν θα ε, υποχωρήσει ως προς τη δική του πολιτική. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει σύνορα. Εάν έχουμε κανόνες δεοντολογίας για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα τεχνολογία, αυτό θα πρέπει να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε επίπεδο όσα στις χώρες όπου θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτανε σε ένα επίπεδο προδιαγραφών έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει ουσιώδης έρευνα σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, τότε θα γίνει κάπου αλλού αυτή η έρευνα. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να τάσεται υπέρ της ανθρωπότητας, να είναι ένα μεγάλο θετικό εγχείρημα και από όσο γνωρίζω η Επιτροπή Απασχόλησης θα γνωμοδοτήσει. Μπορούμε να προτρέξουμε Ξέρουμε τι θα πούν. Η κατάσταση είναι τραγική και πολλοί θα ε, χάσουν τη δουλειά τους. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και 200 ε, χρόνια πριν για την ατμομηχανή. Φυσικά η τεχνολογία καταστρέφει εργασίες αλλά δημιουργεί άλλες και γι' αυτό εμείς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δελεαστικός χώρος για τις επιχειρήσεις και για επενδύσεις. Και αν έτσι προσεγγίσουμε την έκθεση, τότε θα έχουμε καταφέρει πολλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε αυτά που είπατε ως προς το περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο κύριος Μπούζεκ, ε, από το ΕΛΚ ο κύριος Σαουντάργκας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω τα όσα προελέχθησαν από τον εισηγητή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και όλα τα συναφή και νομίζω ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης είναι μια καλή αρχή και μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αλλά αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε διάφορα βασικά μηνύματα όχι σε λεπτομεριακό επίπεδο. έτσι ώστε να μην δούμε ε, ζητήματα ε, τεχνικής υφής, αλλά την ίδια τη γνωμοδότηση. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μεγάλη η παρανόηση της κοινωνίας των ΜΜΕ για το τι συμβαίνει. Τι σημαίνει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το βλέπουμε και στην, ε, στις εκθέσεις που προανέφερε ο εισηγητής. Δεν έχει ε, σχέση με την επιστημονική φαντασία. Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη υπό τη στενή έννοια για συγκεκριμένα καθήκοντα, αλλά πρόκειται για ένα τεράστιο έργο ως προς την αναγνώριση εικόνας και ιδιαίτερα ζητήματα υψηλής πιστότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετάσχει σε τέτοια έρευνα. Αλλά αυτοί οι αλγόριθμοι στην ουσία ε, έχουν ε, διασπαρεί σε πολλές κατευθύνσεις. Θεωρούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη έχει ήδη χάσει, γιατί έχουν γίνει πολλές επενδύσεις ήδη στις ΗΠΑ, στην Κίνα και ούτω καθεξής. Και η Ευρώπη ε, λέγεται ότι δεν θα μπορέσει να συμπαραταχθεί. Εμείς θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένες προτεραιότητες δεν χρειάζεται δηλαδή να ε, τους φτάσουμε σε απόλυτα στοιχεία, αλλά στην ποιότητα. Α, αυτή η τεχνητή ε, νοημοσύνη υπό τη στενή έννοια βασίζεται στα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσεγγίσει το θέμα και ξέρει ποια είναι τα επιμέρους ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, όλα εξαρτώνται από τα εγχώρια στοιχεία, γιατί είναι σαφές ότι το output αυτού του μέσου στην ουσία οδηγεί σε εισρωή στοιχείων, δηλαδή input. Αν έχουμε ένα πρόγραμμα με βάση συγκεκριμένα δεδομένα θα μας δώσει ένα output ενός άλλου πρόγραμμα, σε ένα άλλο πρόγραμμα. Αυτή θα πρέπει να είναι και η νομοθετική μας ε, προσέγγιση, γιατί εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον οποιαδήποτε ε, αλγόριθμο στην Ευρώπη, θα πρέπει να βασιστούμε στα εγχώρια στοιχεία. Ως προς την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, δεν μιλάμε μόνο για τη δεοντολογία και την ε, κακή της ερμηνεία ως προς ε, ζητήματα δήθεν ε, επιστημονικής φαντασίας. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτή τη νοσηρή προσέγγιση. Αυτό δεν έχει να κάνει με νοημοσύνη, αυτό το πρόγραμμα, αυτά τα προγράμματα, γιατί αυτό είναι ένα μέσο που στην ουσία δεν έχει σχέση με τη νοημοσύνη. Είναι ένα μέσο που θα ε, χρησιμοποιείται παντού θα βρίσκεται παντού, στα τραπέζια μας, στο δάπεδο, στα ψυγεία μας, παντού. Δεν πρόκειται για ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Έχει σημασία πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις με βάση τους αλγορίθμους που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή δεν λέμε ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους δεν θα φύγουν οι άνθρωποι από το επίκεντρο. Είναι για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Δηλαδή πολλαπλασιάζουμε την ανθρώπινη εργασία. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω και θα πρέπει να αποστείλουμε αυτό το σαφές μήνυμα. Έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να το προωθήσουμε προς το κοινό μας και στο ε, κοινοβούλιο, το ότι αποφασίσαμε να προωθήσουμε αυτή την έκθεση σημαίνει ότι κάτι θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Εύα Καϊλή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ashley Fox για αυτή την αρχική έκθεση. Πολύ καλό, τον Ashley Fox, με συγχωρείτε, για ε, τα όσα έχει συγγράψει, γιατί με τους χρονικούς περιορισμούς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πάντως εγώ στηρίζω πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και Ενωμένο Βασίλειο. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Δεν είμαστε σίγουροι πως θα μας εγκαταλείψετε. Και δεύτερον, αν δείτε κάθε κράτος μέλος, ακόμα και το Ενωμένο Βασίλειο, δεν είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη ε, στο top 10. Άρα λοιπόν πώς θα ανταγωνιστούμε την Κίνα αν δεν συνεργαστούμε. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι να συνεργαζόμαστε περισσότερο με οποιονδήποτε τρόπο και όπως μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε ε, μια ηγητική θέση όπως έχουμε για την προστασία των δεδομένων, όπως έχουμε για το blockchain, έτσι να κάνουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μόνο στην Ευρώπη έχουμε τη βεβαιότητα πως η χρηματοδότηση θα δοθεί στις ε, επιχειρήσεις που σέβονται τον ιδιωτικό χώρο και την ιδιωτικότητα της ζωής των πολιτών και που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Μπορούμε να το καταφέρουμε, να είμαστε μπροστά, να είμαστε φιλόδοξοι. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, ε, η Κίνα και η παρακολούθηση είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, όχι όμως στην Ευρώπη, όπως επίσης το να βάζουμε σε ε, λίστες τους πολίτες και να τους αποκλείουμε για παράδειγμα από τη δυνατότητα να ασφαλιστούν, να μην επιτρέψουμε τέτοιες διακρίσεις στην Ευρώπη που γίνονται όπως γίνονται στην Κίνα, θα πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να σχεδιαστεί για να έχει και ηθική διάσταση. Ο αλγόριθμος λοιπόν να μιλά και για ηθικά θέματα, όχι μόνο για κέρδος. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να προσφέρει εξηγήσει για τις αποφάσεις που λαμβάνουν αλγόριθμοι με ανθρώπινη ευθύνη και συμφωνώ. Δεν είναι ακριβώς νοημοσύνη, ουσιαστικά πρόκειται για αυτοματοποίηση και αναγνώριση ε, τάσεων. Αλλά θα πρέπει εμείς να θέσουμε τους όρους και το πλαίσιο μέσα στον οποίο θα εξελιχθούν όλα αυτά. Και κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί είναι να αναγνωρίσουμε. Θα χαθούν πολλέ θέσει εργασία, αλλά ακόμα περισσότερε θα δημιουργηθούν. Αυτό εξαρτάται από εμά και τα παιδιά μα ήδη συζητάνε ε, το κατά πόσο θα μπορούν να γίνουν YouTubers ή influencers, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία δεν υπήρχαν. Πρέπει λοιπόν μέσω κωδικοποίησης, μέσω ψηφιακών δεξιοτήτων να τα βοηθήσουμε να το καταφέρουμε. Θέλουμε να εστιάσουμε στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στις νέες ε, θέσεις εργασίας, στην συναισθηματική νοημοσύνη, στην ηθική και βέβαια στις τεχνικές δεξιότητες και όλα αυτά με τρόπους που θα μας ξεκαθαρίσουν ποιος έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί όλα να συμβαίνουν έτσι οι πολίτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να, λάβουν τις να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πάρουν αποφάσεις και πιστεύω πως θα πρέπει να συνεργαστούμε παράλληλα ε, με το σχέδιο δράση της FinTech ε, και να δώσουμε sandbox για τις μικρές εταιρείες έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, τα τοπικά δεδομένα, τα big data, όλα τα ε, δεδομένα που χρειάζονται για να βρουν λύσει και να μην περιορίσουμε την πρόσβαση στα δεδομένα στι πέντε μεγάλε εταιρείε που τα κατέχουν. Θα πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν στοιχεία για να μπορούν ας πούμε, να προλαμβάνουν επιδημίες, ασθένειες, αυτά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η αναταραχή να έχει θετικά αποτελέσματα. Και κάτι που θα συζητήσουμε ακόμα είναι πως η έκθεση αυτή θα ασχοληθεί και με τις μεταφορές. Και σε περίπτωση Ατυχήματο, ποιο είναι υπεύθυνο. Όχι το όχημα βέβαια. Χρειαζόμαστε κέντρα αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη γιατί θα αλλάξει τη ζωή μα. Και θα είναι μια συνεχή διαδικασία. Θα πρέπει επίση να έχουμε και τη δική μας τεχνολογία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να υπερασπιστούμε και να εξασφαλίσουμε τα δεδομένα των συμπολιτών μας ε, τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Είμαστε πολιτικοί. Και αυτό πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Ελπίζω να μην έχουμε καθυστερήσει και ελπίζω πως τουλάχιστον μια έκθεση, ε, θα έχουμε μια έκθεση που θα αποτελεί και παράδειγμα για την υπόλοιπη οικουμένη. Και πως θα την ακολουθήσουν, ε, έτσι όπως εμείς θα την παρουσιάσουμε. Κυρία Νάχτιγκάλ, ευχαριστώ πρόεδρε και να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι το κείμενο λοιπόν είναι καλό και αξίζει τον κόπο και φυσικά πάντα μπορούμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία αλλά να είμαστε προσεκτικοί, να μην το παραφορτώσουμε το κείμενο. Και το κάνουμε χριστουγεννιάτικο βέντρο προσβλέπω και στο σχέδιο δράση για την ε, τεχνητή νοημοσύνη που θα μα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 5 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε πιο πολλές λεπτομέρειε και τροπολογίες που θα ήθελα να καταθέσω θα εστιαστούν ε, στην ανάγκη η τεχνολογία να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη και να υπάρχει πρόσβαση και στην τεχνολογία όπως ορίζεται και στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Και τέλος να προσθέσω ότι είμαστε επιτροπή για τη βιομηχανία. Να μην επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο σε συγκεκριμένους τομείς για την πολιτική, να ενταχθεί αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιομηχανικής στρατηγικής και προσβλέπω στη συνεργασία με τον Άσλη και πάλι για το θέμα αυτό. Grazie. La parola, collega Silichiotis, prego. Εγώ αρχικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Άσλε Φόξ για τη ε, δουλειά που έκανε μέχρι τώρα για την έκθεση και να συμφωνήσω μαζί του ε, σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Ε, έχει δίκιο, δεν μπορούμε να μιλούμε για ότι θα κάνουμε μια σοβαρή δουλειά ε, σε, μέσα από τέτοια ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα, ειδικά τώρα για ένα τόσο ε, ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Είναι γεγονό πω η τεχνολογική εξέλιξη, η ρομποτική και η τεχνική νομοσύνη υπόσχονται πολλά πλεονεκτήματα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ε, ωστόσο, για την ομάδα μα είναι ξεκάθαρο πω για να έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα πρέπει η τεχνική νοημοσύνη, η ρομποτική να αξιοποιηθούν με υπευθυνότητα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αγκών τη κοινωνία, καθώ και για ενίσχυση τη ευημερία, τη ποιότητα ζωή των ανθρώπων, και εδώ πρέπει να είναι ο βασικό στόχο. Ε, και προ αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτήν την νέα δυναμική, την ευκαιρία θα λέγα, που μας δίνεται για να δημιουργηθούν νέε ποιοτικέ και αξιοπρεπείς θέσει εργασία, μέσω της ανάπτυξης τεχνική νομοσύνης. Είναι ένα θέμα που έθεσε και ο συνάδελφο ο Σαντάρκα και σύμφωνο μαζί του. Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε πώ ο τομέας της τεχνικής νομοσύνης τη ρομποτική, θα στηρίξουν το εργατικό δυναμικό που ήδη υπάρχει και αυτό χρειάζεται πραγματικά να υπάρχει και στο υφιστάμενο προσωπικό εκπαίδευση και θα ε, ενισχύσει τις ανθρώπινες δυνατότητες και να δώσουμε νέα όθηση στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Είναι δηλαδή σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ε, τη ρομποτική και την τεχνική νομοσύνη για να καλύψουμε κενά και αδυναμίες που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα πρέπει να σα πω, το είπα και άλλε φορέ, στον Νότο, όπου ε, ο Νότο τη Ευρώπη βρίσκεται σε μια διαδικασία επαναβιομηχανοποίηση και χρειάζεται ακριβώ αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμό. Ε, και είναι ακριβώ σημαντικό να προωθήσουμε την καινοτομία και στον ε, τομέα τη ρομποτική, ώστε να στηρίξουμε αυτή την εκβιομηχανοποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να οθεί και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα το σημαντικό με την τεχνολογική εξέλιξη δεν είναι το μέγεθο τη εταιρεία, αλλά η ποιότητα της, της ε, ε, ε, βιομηχανίας, η ποιότητα δηλαδή της εταιρεία να μπορεί να αξιοποιεί ακριβώ τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών αλλά και της υγείας, όπως σωστά αναφέρει ο εισηγητής, η τεχνική νομοσύνη μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των αγκών των ανθρώπων. Βασική όμως προπόθεση είναι ο έλεγχος, να τον, έχει, τον έλεγχο πάντα να τον έχει ο άνθρωπος ο οποίο να ενεργεί βάσει ηθικών αρχών και με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κλείνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα στοιχείο που απουσιάζει από το προσχέδιο τη έκθεση που ετοίμασε ο συνάδελφο. Πιστεύω πω είναι σημαντικό η Επιτροπή μα να αναφερθεί στην άγκη να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά δεδομένα στην δημιουργία τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ε, εσωμάτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και ιδιαίτερα τη τεχνική νομοσύνη. Ε, προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι και οι τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Άσλεϊ Φόξ για τα όσα μας παρουσίασε. Αυτό το οποίο βρίσκω εγώ πιο ανησυχητικό, ε, γιατί διανύουμε μία περίοδο σχετική ηρεμία. Σκεφτείτε αυτά που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί, τρικυμιώδη. Ε, μιλάμε για δημοσιονομικά θέματα ε, που ε, όπως το Horizon, συγγνώμη, όπως το Europa ε, και τα συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδοτούνται με δις εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα κάναμε με χρόνο ρεκόρ. Οπότε να μην μιλάμε για πιεστικά χρονοδιαγράμματα εδώ, γιατί επαναλαμβάνω το πρωί είδατε τι έγινε. Εξαιρετική δουλειά έκαναν οι συνάδελφοι, αυτό πρέπει να το πω. Και Βεβαίω ε, δεσμεύουμε κονδύλια και είναι δύσκολη η κατάσταση δημοσιονομικά για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη-μέλη, οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναδιατύπωση στο τι σημαίνει και στο ποια είναι η διάστασή τη, γιατί πολλέ φορέ μοιάζει να είναι κάτι καινούριο, κάτι που μόλι εμφανίστηκε, σαν να μην είχαμε τίποτα στο παρελθόν. Αλλά να σας πω πως αποτελεί απλώς μία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι δηλαδή η επεξεργασία δεδομένων που γίνεται από πολύ δυνατούς υπολογιστές. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μόνο που αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ως άνθρωποι όλο και περισσότερα δεδομένα. Και κάθε μέρα έχουμε επεξεργαστές οι οποίοι είναι ακόμα πιο ισχυροί και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε καινούργιες εφαρμογές. Τα λέω αυτά γιατί γιατί θέλω λίγο να χρωματίσω αυτά τα οποία σχολιάζουμε. Δηλαδή, είναι αλήθεια πως αυτή τη στιγμή ξεκινά μια περιπέτεια με ένα κόσμο άγνωστο για μας, που επηρεάζει όλη την οικονομία και που τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω πως θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταφέρουμε. Και για κάποια προβλήματα τα οποία εμφανίζονται και όπου έχουμε μία ε, σταδιακή εξέλιξη που δεν μπορούμε καν να προδικάσουμε προς πού θα πάει. Χρειάζεται να τα σχεδιάσουμε, να κάνουμε κάποια σκέψη. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι πως έχουμε μια σειρά από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε αμέσως με λύσεις που ήδη υπάρχουν. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Το πρόβλημα με τα δεδομένα μας οδηγεί κατευθείαν στο θέμα της συνδεσιμότητας. Μα μόλις ψηφίσαμε κάτι σήμερα το πρωί για να έχουμε κινητά και σταθερά δίκτυα πολύ υψηλή ταχύτητα. Χρειαζόμαστε για παράδειγμα επεξεργαστές πάρα πολύ γρήγορα στην Ευρώπη που δεν έχουμε. Αυτούς τους σούπερ υπερλογιστές. Σήμερα λοιπόν εγκρίναμε ένα πρόγραμμα το Digital Europe, ψηφιακή Ευρώπη, που έχει συγκεκριμένο προπολογισμό για να αγοράσουμε δύο υπερυπολογιστέ στην Ευρώπη που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που πρέπει να πηγαίνουν οι εταιρείε μα στην Ασία ή κάπου αλλού, στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη, στη ΣΥΠΑ, για να ε, βρουν αυτό που χρειάζονται. Αυτά λοιπόν τα έχουμε και στο πρόγραμμα αυτό, το Digital Europe, έχουμε 2,5 δις ευρώ για πουλωτικά προγράμματα για τις εταιρείε και για τις δημόσιες αρχές για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Και μας είπε το Μάιο του 19 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει μια αναθεώρηση για την, ευθύνη, για την οδηγία για την ευθύνη για τα προϊόντα και εκεί θα έχουμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη, το big data, όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε εδώ και τελειώνω. Και θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα κοινωνικά θέματα και για την παιδεία και για την επιμόρφωση, για τα ηθικά ζητήματα που υπάρχουν, για την ευθύνη. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως θα πρέπει την τεχνητή νοημοσύνη να την εφαρμόσουμε αμέσως, μια και είναι πολύ εξελιγμένη. Θα ήθελα να μην μακρηγορείτε, γιατί είναι ε, σημαντικό το θέμα. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Η Τερέζα Κρίφιθ. Γκρίφιν, θα ήθελα να πω με αυτά που είπε η Εύα Καϊλή. Μιλήσατε για ανυπαρξία σύνορων και ξέρω ότι όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην υπάρξουν, να μην ε, σκληρά σύνορα μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας, διότι πολλοί είναι οι άνθρωποι που διαβαίνουν τα σύνορα για να ε, μελετήσουν, να εργαστούν και να επισκεφθούν τις οικογένειές τους. Ζούμε ε, ε, μέσα σε παγκόσμια δεδομένα. Καλή η παγκοσμιοποίηση, αλλά θα πρέπει να γίνει μια σωστή μετάβαση των εργαζομένων και να καταρτήσουμε τα παιδιά μας για εργασία ε, υψηλής δεξιότητας, υψηλών δεξιοτήτων. Άσλεϊ, ε, γίνεται και πολύ μεγάλη έρευνα από τα συνδικάτα που θα πρέπει να λάβεις υπόψη. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο εγώ για ένα λεπτό. Εντάχει, υπάρχει και κάποιος άλλος. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, σας είδα. Είπε κάποιος είναι πολύ αργά, ίσως έχει χάσει η Ευρώπη το παιχνίδι. Άλλοι είπαν ότι είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, των μεταφορών και ούτω καθεξής, δηλαδή να ε, εκμεταλλευτούμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Εμείς ε, έχουμε ως σημείο εκκίνησης τη δεύτερη αυτή προσέγγιση. Όλα αυτά ισχύουν για την Κίνα, τη ΣΥΠΑ, αλλά και ο Καναδάς συμμετέχει σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια. Νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο να εμβαθύνουμε. Όταν συζήτησε ένα think tank είπε ότι ε, εσείς έχετε αιμονή με τους κανόνες και επειδή έχετε αυτή την ιδεολειψία τότε ε, θα αποτελέσετε τροχοπέδι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας όπως ισχύει στη Σιγκαπούρη. Δηλαδή, ε, οι συμβάσεις εκεί είναι πάρα πολύ εύκολες. Μπορεί να είναι και μια διμερή σύμβαση η οποία συντάσσεται και υπογράφεται πολύ εύκολα. Υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί όπως της Οξφόρδης που είπαν ότι πρέπει να ορίσουμε κανόνες για ευθύνη, για ιδιωτικότητα και τη σχέση ανθρώπου με τις μηχανές και αυτός που ορίζει τους κανόνες μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Εάν εμείς λοιπόν ορίσουμε σωστά τους κανόνες, ίσως θα έχουμε ένα καλύτερο χαρτί στη διεθνή σκακέρα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, που έχει σχέση και με τις άλλες μας επιλογές. Μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής Ευρώπης θα πρέπει όμως να έχουμε μία προσέγγιση που να μας διέπει. Εδώ βρίσκεται η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Η κυρία Κούπουλα Νάτρη έχει το λόγο και της δίνω το λόγο. Μετά θα ακούσουμε την Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συζήτηση που γίνεται εδώ σήμερα και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι κάπως ε, με την ε, δομή της δουλειάς μας γιατί είναι πάρα πολύ μικρή η περίοδος που έχουμε και προφανώ πρόκειται για ένα θέμα που επηρεάζει πάρα πολλού τομεί. Ελπίζω λοιπόν και η Επιτροπή Απασχόληση από την οποία προέρχομαι. Τι έχω μάθει από τη Φιλανδία στον τομέα των οικοδομών. Να τη τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν πώς έχει εκπαιδευτεί καθένας και πού μπορεί να βρουν τα πιο καταλάτωμα. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη γενικότερη στρατηγική απασχόληση στον τομέα των οικοδομών. Πραγματικά υπάρχει εφαρμογή παντού και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ε, ένα κατάλογο με τα παραδείγματα, θετικά ή αρνητικά, αλλά να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αρχές για την ανθρώπινη ζωή και κάποιες αρχές ε, από πλευράς της κοινωνίας. Και για να τηρήσουμε αυτέ τι ε, αρχές δεν χρειάζεται να περιορίσουμε και να καταπνίξουμε την καινοτομία στην Ευρώπη. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη σε αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο χαμηλή από τι άλλες χώρες ανταγωνιστικέ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, από τη Γενική Διεύθυνση Connect, κ. Σιλουίντς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Ναι. Μας πιέζει ο χρόνος, αλλά δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Γιατί από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πολλή δουλειά προς την κατεύθυνση αυτή που βλέπουμε και εδώ. Και να πω συγκεκριμένα ότι έγινε πολλή δουλειά σε επίπεδο υψηλών Επιλογνωμόνων για την τεχνική νοημοσύνη προετοίμασαν κάποιε κάποιες γραμμέ που θα δημοσιευτούν το Δεκέμβριο και θα μπουν αυτά στη σχετική πλατφόρμα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου όλοι μπορούν να τα κοιτάξουν. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να κοιτάξω να προσθέσω τα σχόλια που έγιναν για το κείμενο. Και θα ήθελα να πω στο σημείο C μιλάτε για τους κανόνες και τις διαδικασίες. Αυτά είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Αρκετά ξεχωριστά. Οι κανόνες έχουν να κάνουν με την νομοθεσία. Και εδώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες, θα πρέπει να δούμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των κανόνων. Εδώ θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε ενδεχομένω και να χρειαστεί να τροποποιηθούν για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει πραγματικά αντομία Στο σημείο D. Εδώ η διατύπωση ενδεχομένω να είναι κάπω παραπλανητική. Γιατί φαίνεται ότι το σύστημα είναι μεροληπτικό. Ε, να προσέξουμε λίγο. Επίσης αυτό δεν ισχύει για όλα τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη. Δεν βασίζονται όλα σε τέτοια big data. Ενδεχομένω λοιπόν, να πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εγγύηση σε όλε τι περιπτώσει και ενδεχομένω να υπάρχει μεροληψία. Για να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ορισμού αυτή η υποψία για ύπαρξη κατηγορίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Να πούμε επίσης ότι για κάποια καθήκοντα θέλουμε τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε εφαρμογές 3D, τρισδιάστατες και άλλες επικίνδυνες εφαρμογές, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα εργασίας. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε ως δυνατότητα. Και πιστεύουμε επίσης ότι η αυτόνομη οδήγηση τύπου 5 χωρίς μόνη σημαίνει ότι θα αφαιρεθεί και ο οδηγός προφανώς. Να προσέξουμε την διατύπωση. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική στη γυράσκουσα κοινωνία, το 5 και εξής. Εδώ, το σημείο αυτό είναι κρίσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ομοφωνία και συνένεση για τη χρήση τεχνής νοημοσύνης ε, στην φροντίδα, στον τομέα της φροντίδας. Για παράδειγμα, το 2007 που έγινε μια μελέτη, προέκυψε ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αισθάνεται άφολα με την προοπτική να τους ε, παρέχει υπηρεσίε ε, σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων και μόνο 26% των συμμετεχόντων αισθάνονται ασφάλεια. Να προσέξουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά το στόχο που αναφέρεται. Όντω στην Ιαπωνία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είμαι βέβαιη ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσουμε μια τέτοια ρύθμιση όπου 4 στις 5 θα επιλέγουν αυτή την ε, φροντίδα από ρομποτική. Να προσέξουμε. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη των νοσοκόμων να υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη από τη ρομποτική, αλλά και πάλι χρειάζεται αυτή η ανθρώπινη επαφή. Σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, τι ορίζουμε ναι. καλωσορίζουμε αυτή την παράγραφο, γιατί πραγματικά συνάδει με τι αυξημένε επενδύσει που εφαρμόσαμε. Τις αυξήσαμε κατά 70% και καλούμε και τα κρατη και τις εταιρείε να κάνουν το ίδιο. Κάτι που θα θέλαμε να τονίσουμε εδώ, πέρα από τα ρομπότ και την έρευνα θα πρέπει να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη, όπως και το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, να το τονίσουμε αυτό. Το σημείο 7 για την εκπαίδευση. Εγώ θα έλεγα την εκπαίδευση να τη δούμε υπό το ευρύτερο πλαίσιο. Χρειαζόμαστε επίσης να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να γνωρίσουν τι μπορεί να κάνει το σύστημα για αυτούς και πώς μπορεί να βελτιώσει κάποιες ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες και διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική, έχετε παριθμίσει διάφορα θέματα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα. Για παράδειγμα, στον τομέα την αγροφήμων, της περιβαλλοντικής προστασίας και πάλι στον τομέα της υγειονομικής περιθέψης. πολλά παραπάνω μπορεί να γίνουν αυτό ενδεικτικά. Το θέμα της διατολογίας της ηθικής, πολύ κρίσιμο κι αυτό. Ναι, λίγο... Παρακαλώ, ε, τελειώνετε, γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε καθυστερήσει μόνο τα σημεία ουσίας να μας πείτε. Ζητώ συγγνώμη και να κοιτάξω ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα είναι αυτό το θέμα της διαντολογίας, όπου θέλουμε να, να αναφέρουμε ότι αυτό που προτείνεται ουσιαστικά εδώ είναι αυτό που κάνει η ομάδα των εμπειρογνωμών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλή δουλειά λοιπόν θα πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Και θέλουμε να υπάρχει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να δούμε τι έχει κάνει και η ομάδα εδώ. Τελευταίο θέμα και Ελπίζω να μπορέσω να αποστείλω γραπτά τα υπόλοιπα θέματα. Το τελευταίο θέμα που ήθελα να αναφέρω είναι το σημείο 34 για την ε, ορισμό μια task force. Αυτό ακριβώ κάνουμε αυτή τη στιγμή με την ομάδα των υψηλών εμπειρογνωμόνων και με τα κράτη-μέλη και στο συντονισμένο σχέδιο δράση. Θα πρέπει λοιπόν να επεκτείνουμε τη συνεργασία αυτή και με το Κοινοβούλιο. Εδώ θα βάλω ταινία. Σας ευχαριστώ και για τις υποδείξεις. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Ashley Fox και θα ήθελα να πω κατά πόσο είσαστε διαθέσιμοι, θα το πω στον κύριο Μπούζεκ, να έχουμε μία συνάντηση και ακρόαση με αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου και νομίζω ότι μία συζήτηση μαζί τους θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και για εμάς. Γιατί ε, είμαστε διαθέσιμοι από πλευράς Κοινοβουλίου. Ο συνάδελφος Φόξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συνήθως θα απαντούσα στα σχόλια των σχεδόν και στους πέντε ομιλητές και θα τους ευχαριστούσα ξεχωριστά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει. Η δική σας πρόταση που είναι να συναντηθούμε με την ομάδα υψηλού επίπεδου είναι πολύ ε, και αυτό συμβαίνει και ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία και στη Γερμανία όταν περνάνε τέτοια θέματα από τη Βουλή. Και πρέπει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου να έχουμε ε, ε, να έχουμε ψηφίσει και μέχρι 5 Δεκεμβρίου να έχουμε στείλει τροπολογίες. Οπότε πραγματικά είναι πολύ ε, αστείο το ότι μας δίνουν αυτές τις σφιχτές προθεσμίες έχοντας περάσει έξι μήνες συζητώντα σε ποια επιτροπή θα το δώσουν. Θα πρέπει αυτό να είναι ένα δίδαγμα για το μέλλον έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και ακροάσει με τους ε, τα κτλ. Πάντω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συνεργαστούμε με τι άλλε επιτροπές και ελπίζω πω 7 Ιανουαρίου θα έχετε ένα κείμενο στη διάθεσή σα το οποίο θα μπορούν να υπερψηφίσουν οι συνάδελφοι. Ωραία. Ολοκληρώνουμε την άκρος ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Φόξ που μας ανέφερε όλα τα ζητήματα επί της ουσίας. Τώρα, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 6η Δεκεμβρίου στις 12. Από ό,τι κατάλαβα θέλει μια παράταση. Εάν ε, χορηγηθεί θα σας το πω Τερέζα, ένα Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Φόξ για ενδεχόμενη παράταση. Θέλω να με ακούσετε μόνο. Αυτή τη στιγμή η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 6η Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε μετά στις 7 Ιανουαρίου στην Επιτροπή. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς θέλετε να ζητήσετε από τον Μπούζεκ μία παράταση της προθεσμίας, έτσι κατάλαβα Θα ήθελα να αλλάξει την ημερομηνία ψηφοφορίας από τις 7 στις 14 Ιανουαρίου. Άρα 6 Δεκεμβρίου για τις τροπολογίες και μετά θα σας μιλήσουμε, θα σας κοινοποιήσουμε πότε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά τη σήμαση των ελαστικών αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Η κυρία Ντελκαστήλιο θα μας μιλήσει για την έκθεση στη θέση του κυρίου Μπόνη. Uh, uh, uh, Δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να πω δύο λόγια εκ μέρους του. Είναι σύντομο, μην ανησυχείτε. Θέλει να σας ευχαριστήσει όλους γιατί κάνατε πολύ για την έκθεση και συνεισφέρατε πολύ. Η ευρωπαϊκή κινητικότητα θα πρέπει να είναι πιο προσβάσιμη και η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και το η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πιο καθαρή και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται δέσμευση από τα κράτη-μέλη και από τους ενδιαφερόμενους, ε, στηρίζει τις προτάσεις που επιτρέπουν το να φαίνονται οι πληροφορίες για το αν υπάρχουν ε, χιόνια ή ε, πάω ε, στον δρόμο και τα λοιπά και ε, καλωσορίζει τους προθέσεις του, των συναδέλφων να προσφέρουν σε αυτό τις πληροφορίες που θα έχουμε πάνω στα ελαστικά για, τις, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης χρειάζεται μία ε, εμπεριστατωμένη μέθοδος ε, μέτρησης ε, πάνω σε αυτές τις παραμέτρους. Οι έρευνες στον χώρο αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν και αναγνωρίζει πως χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά για την αναγνώριση αυτού της σήμανσης και για το λόγο αυτό χρειάζεται η εισαγωγή μιας νέας σήμανσης Ε, βέβαια μέσα στα πλαίσια των όσων έχουν γίνει στο παρελθόν. Και τέλος θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σχήμα, το, η ίδια σήμανση για, ε, κάποια, για κάποια χαρακτηριστικά ήδη από το τρέχον κανονισμό, για παράδειγμα ε, για τις, για για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα ελαστικά σε υγρές συνθήκες, αλλά και η παραγωγή τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις μας για τη μείωση εκπομπών ε, στην ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ για την εργασία του εισηγητή. Υπάρχουν ε, σημεία τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους ε, την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη συνάντηση σκιωδών για το κείμενο και τις τροπολογίες. Συμφωνώ με όσα προελέχθησαν. Φυσικά υπάρχει και ενεργειακή μετάβαση ε, ε, σε αυτό το τομέα μέσα στα πλαίσια της απομάκρυνσης από τη χρήση άνθρακα. Άρα θα μιλήσω για την αντίσταση κύλησης και άλλα θέματα καινοτομίας με νέες διαδικασίες για τη μείωση αυτή της αντίστασης στην κύληση που αυξάνει την κατανάλωση. Βεβαίως, η σήμανση θα έχουμε το χιλιομετρικό προσδόκιμο, ε, την ασφάλεια και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέξει με κάθε διαφάνεια να έχει τις ε, πληροφορίες για να κάνει αυτή την σημαντική επένδυση. Το θέμα της υγείας και της ανακύκλωσης επίσης έχει σημασία γιατί μας ενδιαφέρει η φθορά των ε, ελαστικών που ε, δημιουργούν, μάλλον διαχέουν μικροπλαστικές ύλες στο οδόστρωμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η επιπρόσθετη μόλυνση που έχει επιπτώσει στην υγεία. Θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες για την ανακυκλωσιμότητα των επισώτρων και ε, σε σχέση με την προμήθεια του καουτσούκ. Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα δράματα που γνωρίσαμε με το Φινικέλεο στο παρελθόν. Είναι δική μας ευθύνη αυτό το θέμα. Αυτό είπε και ο εισηγητής στο μήνυμά του. Να υπάρχει ειδική σήμανση σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσφυσης όταν υπάρχει πάγος στο οδόστρωμα. Τέλος, ως προς τις διάφορες υποκατηγορίες που ζήτησε αλλαγές ο εισηγητής, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Την επόμενη εβδομάδα θα σας πω αν συμφωνώ, γιατί δεν ξέρω αν κατανοώ απόλυτα, τι μας, απόλυτα καλά δηλαδή, σωστά αυτό που μας προτείνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερως που διάφοροι συναδελφοί αναγνωρίζουν την ανάγκη να αναπτυχθεί αυτή η παράμετρος για το χιόνι και τον πάγο στη σήμανση. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό όταν αγοράζει κανείς ένα λάστιχο και πολλές από τις τροπολογίες πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ με την συμφωνία σε ό,τι αφορά να συμπεριλαμβάνονται σταθμισμένοι ταχυδεικτέ για το χιόνι και τον παγό. Να επιστήσω την προσοχή σα για τη χθεσινή ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντο στη γνωμοδότηση για την έκθεση αυτή. Ε, ενέκριναν διάφορε τροπολογίε σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα τη ε, καταμέτρησης καταμέτρηση τη απόστασης, γιατί κάθε χρόνο έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω κακών ε, συνθήκων σε ό,τι αφορά τα λάστιχα και πρόκειται για μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε ό,τι αφορά και τα μικρολαστικά για παράδειγμα. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν ε, διάφορους παράγοντες να αγοράζουμε λάστιχα και να κοιτάξουμε και το θέμα της αντοχής των λάστιχων σε βάθος χρόνου και αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη σήμανση για να υπολογίζεται σωστά το κόστος των επισώτρων. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, το θέμα των μικροπλαστικών είναι βασικό. Και θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν αυτές οι δύο πτυχές στην ε, σήμανση των επισώτρων. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να εμπνευστούμε από αυτά που προτείνουν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος και να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για την προστασία των πολιτών μας. Sì, la Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με κάποια από τα σχόλια που έχουν κάνει οι προλαλήσαντες, αλλά τούτου λεχθέντος πρέπει να σου πω πως τα μικροσωματίδια είναι μεν δυνατόν, είναι, είναι σημαντικά, αλλά ακόμα πιο σημαντικά είναι ο ασφαλής τρόπος ε, ε οδήγησης και τι γίνεται με την κύληση. Κάτι το οποίο είναι ε, πιο σημαντικό από τις εκπομπές μικροσωματιδίων από τα ελαστικά αυτά. Εμείς μπορούμε να κατασκευάσουμε ελαστικά τα οποία δεν πρόκειται να έχουν διαρροή μικροσωματιδίων και να μην έχουν καθόλου εκπομπές. Αν όμως το κάνουμε τότε ε, η αντίσταση κύληση θα είναι μικρότερη με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο ασφαλή. Οπότε τι ακριβώς επιθυμούμε εμείς από ένα ελαστικό. 24 τροπολογίες έχουν υποβληθεί και κάποιες ε, έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, υπό ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί το ελαστικό. Ε, πάνω σε πάγο, για παράδειγμα. Επίσης, τι, πώς χρησιμοποιείται αυτό το ίδιο το ελαστικό σε έναν ε, βρεμένο δρόμο. Και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό και δεν έχει αναφερθεί είναι τι θα συμπεριλαμβάνουμε στη σήμανση. Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε για τα τεχνικά ζητήματα σε άλλη στιγμή, με διαφορετικό κατάλογο. Να δίνουμε ένα link, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε τι λένε όλες αυτές οι πληροφορίες και να προσθέτουμε δεδομένα όσο μα το επιτρέπουν οι τεχνολογικέ εξελίξει, γιατί αν χρησιμοποιείται σε διαφορετικέ επιφάνειε το ίδιο ελαστικό, θα έχει ε, διαφορετική ανθεκτικότητα ε, και διαφορετική ε, τριβή. Και βέβαια όλα αυτά προποθέτουν ότι θα χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο. Μπορούμε να έχουμε νέους μεθόδους δοκιμασίας και τα στοιχεία αυτά να τα δίνουμε όταν κάποιο κλικάρει στο ίντερνετ χωρί να χρειάζεται να κοιτάξει κάθε φορά κάποιο τη σήμανση. Δύσκολο δεν είναι να ε, βρούμε συμφωνία μεταξύ σκιωδών και εισηγητή, οπότε με χαρά περιμένω και εγώ τις συναντήσεις που θα κάνουμε. Um, Ευχαριστώ, Πατρίσια. Και να υποστηρίξω αυτό που είπε ο Γιάκο πριν από λίγο στην παρέμβασή του. Η ασφάλεια και η υγεία είναι κρίσιμη σημασία και εδώ πιστεύουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να φεύγουν το πρωί σπίτι προσδοκώντας ότι θα γυρίσουν ασφαλείς πάλι το βράδυ στην οικογένειά τους. Στην περιφέρειά μου έγινε μια σύγκρουση μετά από ένα φεστιβάλ όπου ο οδηγός και δύο έφηβοι έχασαν τη ζωή, του, τη ζωή τους και προέκυψε στην έρευνα ότι τα λάστιχα ήταν 19 χρόνων στο λεωφορείο αυτό θα πρέπει κάπως να φροντίσουμε να μην μπορούμε να ξεφεύγουν από παραθυράκια οι άνθρωποι και να μπορούμε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και των οδηγών και των υπόλοιπων ε, επιβατών. Και θα ήθελα να μπορέσω να πω στη μητέρα ενός από τους δύο αυτού φίβους ε, που έχασαν το ζωή, Φράνσις Μπουλόι, ονομάζεται ότι κάτι κάναμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για αυτή τη μαρτυρία, Τερέζα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Το λόγο είχε εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Η κυρία Κίσμεν έχει το λόγο. Uh, thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή του κ. Μπόνη, ιδιαίτερα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκτασή του και για την όλη δουλειά που έκαναν και οι υπόλοιποι αξιότιμοι ευρωβουλευτέ που κατέθεσαν ε, τροπολογίε και συνέβαλαν και στη συζήτηση. Καλώ ορίζουμε αυτό που θεωρούμε ότι αποτελεί ευρεία ε, υποστήριξη για την πρόταση αναθεώρηση τη σχετική οδηγία. Να αναφέρω δύο σημεία που επιτρέπετε. Είμαστε ενήμεροι για το θέμα το, της ρεβής και των μικροπλαστικών. Γι' αυτό προτείναμε ρητά να συμπεριληφθούν στην επισήμανση. Αυτή τη στιγμή αναπτυχθεί μια αξιόπιστη διαδικασία δοκιμής για το θέμα της ε, ασφάλειας. Προφανώς και επειδή θέλουμε να εργαστούμε γρήγορα, τάχιστα, από τη στιγμή που θα έχουμε τα αποτελέσματα της δοκιμής, προτείνουμε να γίνουν οι προσθήκες στις ε, με πράξη κατά εξουσιοδότηση. Γιατί αυτή είναι η πιο γρήγορη διαδικασία και προφανώς ε. α, αυτή είναι μια διαδικασία επί της οποίας έχει έλεγχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω, την πρόταση να μην αλλάξουν οι κατηγορίες, να παραμένουν όσοι έχουν στον τρέχοντα κανονισμό. Εδώ να αναφέρουμε το εξή για την ε, κατηγορία άμα, για, τα, για τις υγρές συνθήκες 90% των επισώτρων είναι στις τρεις ε, ανώτατες κατηγορίες. Άρα δεν θεωρούμε ότι αυτό δίνει σωστές πληροφορίες και σωστή καθοδήγηση στον ε, καταναλωτή εδώ πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση. Και σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό θόρυβο, ο γενικό κανονισμό αφαιρεί μια κατηγορία. Άρα, ήδη εδώ δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να επιλύσουμε, αλλάζοντα την κατηγοριοποίηση. Και για την τριβή, όντω δεν είναι τόσο επίγον θέμα αυτό, αλλά 43% των μοντέλων είναι στις ανώτατες τρεις κατηγορίες. Άρα και πάλι υπάρχει συνοστισμός στις πιο υψηλές κατηγορίες και υψηλές ε, μάρκες. Και στο σχετικό οργανισμό πλαίσιο αναφέρθηκε επανειλημμένα το θέμα του να έχει επιλογή ο καταναλωτής και να υπάρχει και κίνητρο ο παραγωγός να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αν ήδη υπάρχει συνοστισμός, αυτό το κίνητρο αφαιρείται. Αυτά, Πρόεδρε, και αν θέλετε άλλες τεχνικές ε, διευκρινήσεις, θα χαρούμε να σας δώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία. Η κυρία Ντεκαστήλιο δεν είναι. Ακούσαμε όμως τη συζήτηση των ουσιοδών, των σχεδόν, με συγχωρείτε. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου του 2019 στην Ήτρε, που θα είναι μία ημέρα ψηφοφοριών, όπως ήταν και η σημερινή. Ναι, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ξαναμιλήσω, αλλά μιλώ με πολύ γενικό και ευρύ τρόπο. Πιστεύω για τους φακέλους κάναμε ένα πολύ μεγάλο ε, μεγάλο λάθος. 14 φάκελοι νομοθετικοί, 17 είναι συγγνώμη, εξαιρετική πίεση και δεν θα είμαστε έτοιμοι. Μας υποχρέωσαν με τέτοιο τρόπο να εργαστούμε και οι εκθέσεις ε, με πάνω από 4.000 τροπολογίες σήμερα το πρωί, κανείς δεν τις ξέρει και δεν τις γνωρίζει. Ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα που προσπαθεί να μας, που προσπαθεί να μας παγιδεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έπρεπε να ξυπνήσουν έξι μήνες πριν το τέλος. Ας ηρεμήσουμε. Ας ηρεμήσουμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην κάνουμε ό,τι λάχει. Μάρτιν, έχεις ε, δίκιο. Είναι μια συζήτηση ε, που θα πρέπει να απασχολήσει τους συντονιστές. Και εγώ θεωρώ ότι με κατακλίζουν αυτά τα θέματα και θεωρώ ότι δεν μπαίνω στην ουσία όπως θα έπρεπε ε, με βάση, γιατί στην ουσία βομβαρδιζόμαστε από παντού. Θα πρέπει λοιπόν να το δουν οι συντονιστές και θα το δουν το ζήτημα με τον Πρόεδρο. Παίρναμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στο τομέα της ε, πυρηνικής ασφάλειας μέσα στα πλαίσια του Μηχανισμού Γειτονίας και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της ε, Σύνθηκη Ευρατόμ. Ο κύριος Ούρουτσεφ είναι ο εισηγητής, τον οποίο δίνω και το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας πω καταρχήν πως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έστειλαν τροπολογίες και να ευχαριστήσω κυρίως τους σκιώδεις μας για το γεγονός ότι έλαβαν με πολύ παραγωγικό τρόπο ε, μέρος στη δουλειά που κάναμε και να σας πω το οργαλείο αυτό θέλει να εξασφαλίσει την πυρηνική ασφάλεια στις τρίτες χώρες. Είναι ο μηχανισμός μας για να έχουμε την πυρηνική ασφάλεια παγκοσμίω και να μπορούμε να ανοιχνεύουμε ε, προβλήματα στις ισχύουσες ε, ρυθμίσεις ασφαλείας, να τα διορθώνουμε και να μην ε, επιτρέπουμε να συμβαίνουν πυρηνικά ατυχήματα. Θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες και θα τους ε, στηρίξουμε όχι έτσι γενικά αλλά με συγκεκριμένο τρόπο βασιζόμενοι στα κεκτημένα της κοινότητας Ευρατόμ και με την πραγματογνωμοσύνη που έχουμε στην προστασία από τη ραδιενέργεια στο χώρο τον πυρηνικό. Μετά από την πολύ καρποφόρο ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα με τους σκιώδεις, ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στα εξή. Καταρχήν, διαφάνεια. Διαφάνεια στις αποφάσεις για τα πυρηνικά που λαμβάνονται από τρίτες χώρες. Ήταν ένα, μέρο, ένα μέτρο το οποίο ανησυχεί πολλούς συναδέλφους γιατί θεωρούν πως το επίπεδο διαφάνειας και το πόσο ανοιχτές είναι οι αρχές σε τρίτες χώρες σε σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης για θέματα πυρηνικά είναι ένα θέμα στο οποίο καλό είναι να βελτιωθούμε. Και κυρίως για όσους είναι στην άμεση γειτονία μας. Και γι' αυτό πιστεύω πως θα πρέπει τα θέματα για τη διαφάνεια να φύγουν από τα εκτιμώντα και να μπουν στο διατακτικό και στηρίζω τι σχετικέ τροπολογίε. Τούτου λεχθέντο, α έχουμε ένα ξεχωριστό άρθρο στον κανονισμό που να στηρίζει την ανάγκη της διαφάνειας σύμφωνα και με την κείμενη ε, νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη πως είναι πολύ ε, ευαίσθητες αυτές οι πληροφορίες. Το δεύτερο. Ε, για τη συνεργασία στα θέματα πυρηνική ασφάλειας. Στηρίζω του συναδέλφους οι οποίοι προτείνουν να επαναγκαταστήσουμε στο νέο κανονισμό ένα κομμάτι από αυτά τα συνολικά κριτήρια που ε, ασφαλίζονται, που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα, στον τρέχοντα κανονισμό για την συνεργασία για την πυρηνική ασφάλεια και που έχουμε ε, ήδη ενισχύει. Έτσι ώστε να έχουμε αμοιβαία αλληλοκατανόηση για το τι σημαίνει αυτό το εργαλείο ε, σε επίπεδο ενδιαφερομένο. Τώρα, για την αιρεσιμότητα. Να σας πω πως κατά τη γνώμη μου οι προϋποθέσεις που ζητούν οι συνάλφοι να εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο δεν είναι αρκετά ισορροπημένες. Και αν τις εγκρίνουμε θα αποθαρρύνουμε πολλούς από το να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Θέλουμε πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, αλλά αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές πολλοί δικαιούχοι θα αποκλειστούν γιατί θα είναι από χώρε όπου οι αρχές αυτές δεν γίνονται σεβαστές. Είναι προβληματικές. Υπάρχει κι άλλο ένα όργανο διεθνούς συνεργασίας που έχει τους ίδιους στόχους που έχουμε κι εμείς. Εκδημοκρατισμός, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ το κομμάτι της πυρηνικής ασφάλειας είναι ε, κάτι το οποίο βλέπουμε συνδυαστικά. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε την ευελιξία που θα μας επιτρέπει να λύνουμε αυτά τα θέματα στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε με τις τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό αυτά να τα ξαναδούμε και να δούμε πώς μπορούμε να χαλαρώσουμε αυτά τα κριτήρια έτσι ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματά μας. Τώρα, υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία δεν συμφωνούμε τόσο είχαμε στο παρελθόν. Τι γίνεται με κοινότητες που είναι σε φάση μεταβατική. Μπορούμε να στηρίσουμε εκεί τη διαχείριση της μέτρησης της ραδιενέργειας, για παράδειγμα. Και όλα αυτά εμπίπτουν στο εργαλείο μας. Νομική βάση, εκεί έχουμε κάποιες ενστάσεις. Ζήτησα νομική γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία και σας έχει σταλεί. Η συνθήκη πάντως Ευρατών είναι όντως το, η κατάλληλη βάση, νομική βάση για το εργαλείο μας. Και εδώ θα το κλείσω. Ήσασταν πολύ διεξοδικός παρά τη διακοπή σας. Λοιπόν, τώρα αρχίζουμε με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Τέλιτσκα. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Θα ήθελα να θίξω ένα μόνο θέμα, αλλά θα πρέπει να πω ότι οι συμβαστικές τροπολογίες εντάχει γιατί ήμουνα σε έναν τριμερή χτες το βράδυ μέχρι αργά και έδωσα και τελική μορφή στο ΣΕΦ, στο Συνδέοντα στην Ευρώπη, που θα μας απασχολήσει αύριο. Αλλά συμφωνώ στα επτά σημεία που είπε ο εισηγητής. Το θέμα είναι η πρόθεση μεταξύ με, με, μερικών συναδέλφων να θέσουν το θέμα της επικουρικότητας όπως ε, πρότειναν και για τα ανθρώπινα δικαιώματα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια συμφωνία με βάση ένα διαφορετικό άρθρο όπου θα γίνουν παραχωρήσεις και θα πρέπει να υπάρχει επικουρικότητα όπως ίσχυσε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε για τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας στις χώρες που δεν απέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση γείτονες χώρες και άλλα βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν νομίζω ότι η στεναρή επικουρικότητα θα προωθήσει την ασφάλεια ή τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί μιλάμε για χώρες που δεν θέλουν καν να μπουν σε διάλογο για την πυρηνική ασφάλεια γιατί είναι ευαίσθητο θέμα για αυτές. Και γι' αυτό δεν έχει νόημα να επιμένουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι η προσέγγιση της έκθεσης είναι πολύ σωστή ως προς τη νομική γνωμοδότηση. Πάντα βασιζόμαστε στο άρθρο 203 της Ευρατών. Και αυτό ακριβώς μας είπε και η νομική υπηρεσία. Θα ήθελα να το ξαναδούν οι συνάδελφοι που διαφωνούν. Νομίζω ότι θα δώσουμε τελική μορφή στις συμβαστικές με τον εισηγητή πολύ σύντομα. Χόλιτσεκ. Ευχαριστώ. Και χαίρομαι που ακούω ότι ο συναδελφός μου προσπαθεί να επικεντρωθεί σε αυτό που πραγματικά έχουν σημασία. Και όχι τόσο στους ε, όρους και στους τρόπους που ενδεχομένω να συνεργαστούμε ή όχι με τις χώρες αυτές. Θα πρέπει καταρχά να δούμε λοιπόν ε, τι κάνουμε κι εμείς. Έχουμε πολλά να πούμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά που είναι αντίθετα με την, ε, το χάρτη των δικαιωμάτων, με τον ΟΓΙΑ κτλ. Να δούμε λοιπόν. Έχουμε πάντα τη διεθνή υπηρεσία, η οποία πάντα θα πρέπει να την συμβουλευόμαστε. Να το έχουμε υπόψη μας. Η Ευρατόμ θα πρέπει να υπάρχει μια ανατοτή αρχή για την συνεργασία, για την παροχή υποστήριξης. Αυτή θα πρέπει να είναι τελική αρχή που θα μας βοηθά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μπει στο κείμενο. Αν θέλουμε να κινηθούμε σε τομείς όπου δεν ε, έχουμε παρέμβαση του ΙΚΑΟ, θα φανεί λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει από μόνη της να επιλύσει θέματα τα οποία ο υπόλοιπο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να τα επιλύσει καλό θα ήταν να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου συνεργασία στις γειτονικέ χώρες. Αν θέλουμε όμως να καταστούν όλα αυτά ελκυστικά, θα πρέπει να σκεφτούμε καλά το πώς θα γίνει ακριβώς η διαδικασία αυτή. Έγινε σε χάρα τον εισηγητή και σύμφωνο και με τον κύριο Τελετσικά, ε, κατά εξαίρεση, ο οποίος δεν είναι όμως πλέον εδώ και σας ευχαριστώ. Ο κύριος... Όχι, κύριε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας διακόψω μόνο για μία στιγμή. Όχι, όχι, εγώ έκανα λάθος, το λόγο έχει ο κύριος ε, Μάγερ. Ευχαριστώ και θα προσπαθώ να θέσω τα θέματα αυτά στο πλαίσιο του και να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου θέσατε. Να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τη δουλειά που έκαναν για ένα εργαλείο το οποίο δεν είναι αρκετά εύκολο να το κατανοήσουμε, είναι πολύ τεχνικό. Αποτελεί ένα παράθυρο το οποίο ενδεχομένω να είναι λίγο πιο ασαφές αλλά πολύ σημαντικό παρόλα αυτά. Να, σας ευχαριστήσω για τις τροπολογίες σας που μας βοήθησαν πολύ να συλλογιστούμε κι εμείς σε ό,τι αφορά το νέο αυτό πρόγραμμα. Το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια μια δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ξεκίνησε την δεκαετία του 90 μετά το USS και προφανώς και μετά από το φρικτό ατύχημα του Τσέρνομπελ. Από τότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βοηθά τις χώρες της γειτονίας και της ε, πρώην Σοβιετικής Ένωσης να βελτιώνουν την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών τους για να μην υπάρξει δεύτερο Τσέρνομπιλ. Σε όλα τα εργαλεία τα οποία έκτοτε έχουν δημιουργηθεί έχουμε καλέσει και παρατραίνει πολλά κρατημέλη, πολλά αλλά και τρίτε χώρε να κλείσουν εργοστάσια τα οποία θεωρούσαμε επικίνδυνα γιατί δεν ήταν στο επίπεδο ασφαλείας που θα έπρεπε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Από το 2007 οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συνεργασία μας με τη Ρωσία μας οδήγησαν να πιστέψουμε ότι όλη αυτή η εμπειρία που έχουμε συλλέξει με πρώην Σοβιετικέ χώρες θα ήταν χρήσιμη σε χώρε οι οποίε ήθελαν να βελτιώσουν ε, την παραγωγή πυρηνική ενέργεια ή να ξεκινήσουν την παραγωγή πυρηνική ενέργεια. Όταν μιλώ για πυρηνική ενέργεια ε, εννοώ ε, και άλλε δραστηριότητε πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει και το σύστημα των αντιδραστήρων, τη έρευνα, δεν είναι μόνο δηλαδή μόνο οι σταθμοί. Ε, όλα αυτά είναι εξίσου επικίνδυνα παρά το γεγονό ότι υπάρχει διαφορά ένταση. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε και με τέτοιε εγκαταστάσει, οι οποίε κυρίω βρίσκονται σε λιγότερο αναπτυγμένε χώρε αλλά και στην Αφρική. Οι εγκαταστάσει λοιπόν αυτέ είναι χαμηλή ασφάλεια, είναι υψηλού κινδύνου για του οποίου τίθεται θέμα και ασφάλεια ασφάλεια ε, που δεν αποτελεί το αντικείμενο των εργαλείων και των μηχανισμών που ζητάμε σήμερα, αλλά των ε, εργαλείων και μηχανισμών που αποσκοπούν στην ειρήνη και στη θεωροποίηση, τα οποία επίσης υπάρχουν ως μηχανισμοί. Για την νομική βάση τώρα, νομίζω ότι το έχετε πλήσει το θέμα αυτό μεταξύ σας. Να σας πω όμως ότι αυτό το εργαλείο δεν θα ασχολείται μόνο με τις ε, δραστηριότητε ε, Υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα, ασφάλιση κτηρίων. Αυτό μπορεί να γίνει και από άλλα μέσα, για παράδειγμα, τα εργαλεία για την γειτονία. Και αυτά τα ε, μέσα, λοιπόν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήδη σήμερα για να γίνουν πολλές τέτοιες δραστηριότητε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την Κεντρική Ασία και την ε, χρήση κτηρίων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και για τις ε, σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας για τα θέματα αιρεσιμότητας. Πρόκειται προφανώς για ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας. Παρατηρήσαμε ότι στις χώρες όπου η αιρεσιμότητα μπορούσε να παίξει ρόλο και αυτές είναι κυρίως οι χώρες όπου υπάρχει θέμα ασφάλεια και ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Το Ιράν το πρινικό πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα είναι αυτό που βασίζεται στη συμφωνία του 2015, βάσει του οποίου οι Ιρανοί κατηγορούνται ότι δεν ε, ότι δεν πληρούν ε, τα, τις προδιαγραφές για δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και βάσει αυτής της συμφωνίας οι Ιρανοί δέχθηκαν να ανοίξουν τις πόρτες τους και να γίνουν ε, ελέγχει. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα καλά παράδειγμα το πώς μπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκε σε διάφορες χώρες. Δεν μπορούμε φυσικό να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα σε όλες τις χώρες. Μιλήσατε επίσης για την ευελιξία. Την άκουσα αυτή τη λέξη. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε αυτή την ευελιξία. Γιατί είναι απολύτως ε, κρίσιμη ο κόσμο τη πυρηνική ενέργεια και τεχνολογία εξελίσσονται τόσο γρήγορα και όλε αυτέ οι εφαρμογέ τη στρατηγική και τη πυρηνική ενέργεια εξελίσσονται τόσο γρήγορα που πρέπει και εμεί να τι ακολουθήσουμε. Δεν μπορούμε. Ε, επτά χρόνια είναι μεγάλη περίοδο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο τέλο τη περίοδο αυτή. Και να σα υπενθυμίσω ότι τα βασικά μέσα και τα εργαλεία αυτά και τα μέσα ασχολούνται βασικά με την ασφάλεια των ε, χώρων σε ό,τι αφορά την παροχή υποστηρίξη ε, και καθοδήγηση για τους ε, υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο θέμα σοβαρά, όπως ε, προέκυψε αυτό στην Αρμανία ή σε πυρηνικές εγκαταστάσεις σε χώρες προσχώρησης όπως η σε πρινικες εγκαταστασεις σε χωρες προσχωρησης οπως η σερβια για δραστήρες έρευνας. Εκεί τύφεται δηλαδή θέμα λειτουργίας πιο πολύ των αντιδραστήρων Ευχαριστούμε ιδιαίτερα του ε, βουλευτές για τα θέματα τα οποία υπογράμμισαν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Όντω, για εμά, όπω και για όλο τον κόσμο, η αξιολόγηση του αντικτύπου των προγραμμάτων που έχουμε θέσει σε εφαρμογή είναι βασική. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε σωστούς δείκτες, καταρχάς για να ξέρουμε πώς έχει κατάσταση στην κάθε χώρα, στην εκάστοτε χώρα, όπου βρίσκεται η εγκατάσταση την οποία εξετάζουμε και κατά δεύτερον για να αξιολογήσουμε κατά πόσον όλα τα προγράμματά μας βελτίωσαν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. και μεταξύ άλλων και τις ικανότητες επιθεώρησης από τις εθνικές αρχές του κράτους μέλους. Να διαπιστώσουμε λοιπόν αν υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Είναι ένα είδος ε, stress test ε, για τις συζητήσεις αυτές που γίνονται σχετικά με το ποιο θα κάνει την επιθεώρηση προκειμένου να είναι σωστό το stress test. Εμείς προφανώς δεν μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το αποφασίσουμε αυτό, αλλά εμείς μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη στις εθνικές ε, υπηρεσίες ασφάλειας σε ό,τι αφορά την ε, διεξαγωγή των stress test και να συνεργαστούμε με το Διεθνή Οργανισμό στη Βιέννη, γιατί είναι δική τους δουλειά και δικό του καθήκον να επιθερήσουν την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία, ότι ναι, είναι επιτακτική ανάγκη, είναι και πρέπει να συνεργαστούμε με τις άλλες ε, υπηρεσίες. Η πρώτη είναι προφανώς η υπηρεσία στη Βιέννη, αλλά υπάρχουν και άλλες περιφερειακές οργανώσεις στην Ασία, την Κεντρική Ασία, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι γίνεται πρόοδος και σε περιφερειακό επίπεδο και ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών. Γιατί από ό,τι ξέρετε καλά και όπω είπατε, ε, δεν είναι αντίθετο θέμα εθνικών συνόρων για τη ραδιενέργεια και για τα ατυχήματα. Ζητούν βίζα. Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα. Θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών πυρηνικών μέσων με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων και το μέσο σταθεροποίησης, γιατί υπάρχει κοινή, κοινό στόχο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των υλικών, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Όλα λοιπόν που έχουν να κάνουν με δικλείδες ασφαλείας είναι θέματα τα οποία είναι πολύ κοντινά και άρα η συνεργασία είναι σε καθημερινό επίπεδο θα έλεγα. Και το προωθούμε αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να προωθούνται όλα αυτά με σωστό τρόπο και αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα γιατί το θέμα είναι εξόχως τεχνικό και Ζητώ συγγνώμη αν παρόλα αυτά με ακρηγόρησα. Ε, ναι, Σας έδωσα χρόνο γιατί το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάιερ που είναι σκιώδης από το EFTD. Σας ευχαριστώ. Μου ζητήσατε μόλις έμπαινα αν ήθελα το λόγο. Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε φτάσει στο σημείο αυτό για το οποίο κελτά. άλλωστε. Είπα όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να πάρω το λόγο σας. Ευχαριστώ που μου το δίνετε λοιπόν. Να ευχαριστήσω λοιπόν πολύ τον εισηγητή για τη συνεργασία, για τις ε, συναντήσεις που είχαμε ως τώρα. Είμαστε σε καλό δρόμο και νομίζω ότι θα βρούμε καλούς συμβιβασμού που θα ενισχύσουν ακόμα περαιτέρω τη συμφωνία σε τελική ανάλυση και θα συμπεριλάβουν και τη διάσταση του πολίτη, γιατί για η πολιτική μου ομάδα είναι σημαντικό να διευκρινιστεί στη βασική νομική πράξη ότι μιλάμε για πολιτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και για τη χρήση της ατομικής ενέργειας δεν θέλουμε να την προωθήσουμε έμεσα ή άμεσα. Θέλουμε η προστασία των πολιτών από κινδύνους ατομικής ακτινοβολίας να τονιστούν ιδιαίτερους και να υπάρχει και μεγαλύτερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά την κατάσταση της ασφάλειας των εκάστοτε καταστάσεων στην κάθε χώρα. Γι' αυτό λοιπόν προτείναμε ένα άρθρο το οποίο θα φροντίσει για μεγαλύτερη διαφάνεια τίθεται και θέμα συμπληρωματικότητα με διεθνείς οργανισμούς και συμβάσει οι οποίε θα πρέπει επίση να λεφτούν υπόψη στη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση το ακούσαμε αυτό. Ελπίζουμε το διεθνέ καθεστώ για την πυρηνική ασφάλεια να καταστεί πιο ομοιογενέ και ενισχυμένων. Σε αυτό συγκαταλέγεται και η αρχή της μη διάδοση, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί. Στα θέματα τη ρεσιμότητα. συμφωνώ με αυτά που είπε μόλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ. δεν είμαστε πάντα αντιμετωπισμένοι με δημοκρατίες οι οποίε λειτουργούν όπως θα θέλαμε. Και Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά με υπερβολική ρεσιμότητα σε ό,τι αφορά τι διατάξει ε, κράτου δικαίου, γιατί τα πράγματα στους πυρηνικούς ε, σταθμούς που προχωρούν ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κράτος δικαίου ή όχι. Το θέμα λοιπόν είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες, τον κόσμο, όχι μόνο στην εκάστοτε χώρα, αλλά και στις γειτονικές χώρες, σε όλη την περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει διάλογος με τις χώρες αυτές. Να υποστηρίζεται αυτό από το πρόγραμμα, αλλά να μην ε, διαμορφώσουμε τους όρους με τέτοιο τρόπο. Και αναφέρατε το παράδειγμα του Ιράν. Ε, είχαμε και τον κατάλογο με τα ειδικά μέτρα και τις αναφορές ε, για καθοδήγηση και θα το τηρήσουμε αυτό ως κατευθυντήρια γραμμή για τις περαιτέρω μας εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ούρτσεφ για τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι όλα τα προβληματικά σημεία αποσαφηνίστηκαν. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Κατά τη συνάντηση των σκιωδών συζητήσαμε οκτώ προτάσεις ε, συμβιβασμού και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και θα ήθελα να επιταχύνουν τις ε, τελικές σκέψεις για τις τροπολογίες και να μας πούν ποιες υποστηρίζουν. γιατί θα ψηφίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή. Ωραία. Μας δώσατε και την προθεσμία. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να αρχίσουμε με το workshop που έχει σχέση με το Brexit και τις επιπτώσεις ε, στο πρόγραμμα ορίζον με τους εμπειρογνώμονες που θα ήθελα να έρθουν εδώ. E Και θα σας τους παρουσιάσω. Έχουμε μία ώρα για αυτό το ε, σεμινάριο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα. Θα ήθελα να έρθετε εδώ ο πρώτος ή η πρώτη ομιλήτρια. Βλέπω ότι είναι τρεις κυρίες. Με μεγάλη χαρά. Έντονη γυναικεία παρουσία λοιπόν. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την κυρία Φέγγελερς που θα μας μιλήσει για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του Brexit στο πρόγραμμα Horizon. Yes, uh, good afternoon everybody and uh, thank you for inviting us here to come about To come and talk about the impact of... Θα σας μιλήσω για τις επιπτώσεις του Brexit στο πρόγραμμα Ορίζοντας είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για το ε, Brexit γιατί υπάρχει μεγάλη ε, αμφιβολία και ανησυχίες για το τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας δείξω πώς ε, το πρόγραμμα Horizon Europe θα πρέπει να προχωρήσει ιδεατά όταν θα είμαστε, θα είμαστε μια Ευρώπη των 27 μετά το Brexit. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω ορισμένα στοιχεία ε, μορφή εισήγησης για να δούμε πώς ε, η παγκόσμια κοινότητα έρευνας εξελίσσεται και πώς θα εξελιχθεί το πρόγραμμα Horizon Europe. Δηλαδή η παγκόσμια ε, έρευνα γίνεται πολυπολική με ηγέτιδα της ΙΠΑ αλλά και η Κίνα είναι ένα ανερχόμενο αστέρι. Και αυτό που έχει σημασία να λάβουμε υπόψη ότι και η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος πόλος και από ποιοτική πλευρά και από πλευρά αριστείας. Αλλά βέβαια είμαστε λιγότερο δυναμικοί σε σχέση με την Κίνα και μέσα στα πλαίσια του παγκόσμιου, της παγκόσμιας ε, κοινότητας έρευνας θα πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην Ευρώπη στο μέλλον. Και μέσα στα πλαίσια της ε, πολυπολικής κοινότητας έρευνας θα πρέπει να δούμε πώς θα αναπτυχθεί η αριστεία γιατί το επιστημονικό ταλέντο προσελκύει τους καλύτερους όπου και να βρίσκονται για να χτίσουμε αυτή την αριστεία και να προσελκύσουμε τους ερευνητές. Ένας άλλο σημαντικός μηχανισμός σχετίζεται με την επιστημονική συνεργασία με τα καλύτερα ταλέντα όπου και να βρίσκονται στον κόσμο. Όχι μόνο να τους προσελκύσουμε, αλλά και να συνεργαστούμε μαζί τους όπου και να βρίσκονται στον κόσμο. Έτσι θα οικοδομηθεί η αριστεία. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολυπολική κοινότητα και αν θέλουμε να είμαστε ηγέτιδα δύναμη θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Γιατί αυτό σχετίζεται και με την αριστεία, αλλά και πέραν αυτής. Έχει σημασία που βρίσκονται αυτοί οι επιστημονικοί πόλοι, πώς θα τους εντοπίσει η βιομηχανία για να δημιουργηθούν οι νέες καινοτομίες και η προστιθέμενη αξία. Επίσης, στα πλαίσια της πολυπολικής επιστημονικής κοινότητας, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ανοιχτή και να ε, δελεάσει τα ταλέντα, να τα προσελκύσει μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου, μέσα στα πλαίσια των ανοιχτών οριζόντων και να δούμε ποιες είναι και οι επιπτώσεις με ένα παίκτη λιγότερο μέσα στα πλαίσια του Horizon Europe. Αυτά θέλω να σας πω με αριθμητικά στοιχεία και γραφικές παραστάσεις. Πρώτον βλέπουμε πώς η νέα γεωγραφία καταρτίζεται. Αν δείτε λοιπόν την επιστήμη παγκοσμίως βλέπετε ποια είναι η θέση της Ευρώπης με ή χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπετε ότι η Ευρώπη έχει πολλά δημοσιευμένα πονήματα, γιατί αυτό είναι μια μονάδα μέτρησης. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις η Ευρώπη δεν τα έχει καταφέρει και πολύ άσχημα ε, είμαστε παρόμοια δύναμη σχεδόν με τη ΣΥΠΑ που είναι στην εμπροστοφυλακή. Αν δείτε τη ε, σύγκριση διαχρονικά βλέπετε την αναδυόμενη Κίνα και γι' αυτό ακριβώς και οι άλλοι πόλοι θα πρέπει να τις δώσουν χώρο και ιδιαίτερα η Δύση για να αναπτυχθεί η Κίνα. Άρα παραχωρεί χώρο ή ΙΠΑ. Είναι και η μεγαλύτερη χώρα που έχει και τις καλύτερες δημοσιεύσεις. Η Ευρώπη επίσης είναι ένας βασικός παίκτης σε επίπεδο αριστείας και κατάφερε να κρατήσει τη θέση της διαχρονικά. Δηλαδή δηλαδή δίνει λιγότερο από τις ΗΠΑ, αλλά ε, δεν παραχωρεί τόσο πολύ χώρο στην Κίνα. Έχουμε λοιπόν τις ΕΠΑ Καταρχήν, φυσικά έκανα τους υπολογισμούς με και χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα χάσουμε πολλά βεβαίως χωρίς την, χωρίς την παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θεωρώ ότι άλλες χώρες έχουν παρισφρήσει στο μεταξύ. Άρα η Ευρώπη είναι ένας πόλος δίπλα στους άλλους. Μιλάμε λοιπόν για έναν πολυπολικό κόσμο και φυσικά ο ρόλος της Κίνας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μπορεί να επαυξηθεί στο μέλλον και οι ΙΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν τη θέση τους. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν πώς χτίζουμε αυτή τη θέση αριστείας, πώς έχουμε ε, αριστεία στην επιστήμη της Ευρώπης, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικοί μηχανισμοί που επιτρέπουν στα κράτη να παραμείνουν στην αριστεία καταρχήν να δελεάσουν ταλέντα από, από όπου και να βρίσκονται, άρα η κινητικότητα ταλέντων έχει μεγάλη σημασία και αριστερά βλέπετε ε, πώς έχει ο ακαδημαϊκός κόσμος στην Ευρώπη. Η Ελβετία έχει μεγάλη επιρροή στο δίκτυο. Δυστυχώς οι διερμηνείς δεν διαθέτουν αυτή την παρουσίαση. Έχουμε λοιπόν και έναν ανοιχτό πόλο με την Γερμανία, τη Γαλλία, που είναι μεγαλύτερες χώρες, που δεν είναι τόσο ανοιχτές. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι αυτό το άνοιγμα επιτρέπει την οικοδόμηση της αριστείας. Αυτό βλέπετε στην δεξιά πλευρά. Δηλαδή, αυτοί που προσελκύουμε έχουν ένα σκορ πάνω από το μέσο όρο. Και αυτό έχει σημασία. Αν δείτε τις είπα, η ίπα έχει το, την υψηλότερη βαθμολογία, αλλά βλέπετε ότι ο τύπος έρευνας ε, είναι ε, υψηλότερος. Άρα είναι στην εμπροστοφυλακή γιατί μπορεί να προσελκύσει καλύτερα ταλέντα γιατί προσελκύει τους καλύτερους και καταλαβαίνετε ότι είναι ένας κύκλος, δηλαδή προσελκύει τους καλύτερους γιατί είναι και οι καλύτεροι. Αυτοί που φεύγουν είναι καλοί, αλλά όχι τόσο καλοί από αυτούς που προσελκύουμε και παραμένουν. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Στην Ελβετία έχουμε ένα καλό παράδειγμα βλέπουμε ότι προσελκύουν ταλέντα, αλλά τα καλύτερα ταλέντα. Δηλαδή το ποσοστό είναι υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων στην ε, Ελβετία. Το ίδιο ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει υψηλό επίπεδο αριστείας διότι προσελκύει τους καλύτερους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανοιχτό ορίζοντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υποβαθμιστεί η Ευρώπη. Η Κίνα είναι ένα άλλο παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εισρωή, αλλά και πολύ επανα πατριστέντες που είναι καλύτεροι από το μέσο όρο, αλλά όχι τόσο καλοί όπως τα ταλέντα τον είπα. Βλέπετε στην ε, Κίνα αυτοί που φεύγουν για να πάνε αλλού ε, παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό. Άρα η Κίνα χτίζει την αριστεία της στέλνοντας τα καλύτερα ταλέντα ελπίζοντας ότι θα επαναπατριστούν. Αυτός είναι ο σημαντικός ε, παράγων και φυσικά οι περισσότεροι ερευνητές από την Κίνα θα πάνε στη ΣΥΠΑ. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη πορεία μεταξύ Κίνα-ΣΥΠΑ. Αυτό αυτός είναι ένας ε, τρόπος ε, να χτίζει κανείς αριστεία, να προσελκύει τα ταλέντα και τη δυνατότητα να κρατήσετε τα ταλέντα στην χώρα ή στις χώρες. Επίσης έχει σημασία η συνεργασία με άλλα ταλέντα. Όχι δηλαδή να προσελκύουμε, αλλά να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους όπου και να βρίσκονται. Η διεθνή συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα επίσης που προαγάγει την αριστεία. Ξέρουμε ότι υπάρχει διεθνή συνεργασία και η διεθνή συνεργασία έχει υψηλότερη ποιότητα, δηλαδή αποτελεί προστιθέμενη αξία. Ε, κάτω βλέπετε ε, συνεργασία μεταξύ Γερμανίας, Βασιλείου και Γαλλίας σε σχέση με την βιομετρική. Βλέπετε λοιπόν τις δημοσιεύσεις ε, μεταξύ Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου Έχουμε λοιπόν ε, επτά φορές περισσότερες υψηλότερες δημοσιεύσεις από τις δύο αυτές χώρες. Άρα η αριστεία είναι πολύ σημαντική για να είναι κανείς στην εμπροστοφύλακη και θα πρέπει να χτίζεται μέσα στα πλαίσια των ανοιχτών οριζόντων για να μπορεί κανείς να συνεργάζεται. Οπότε προκύπτει το εξή ερώτημα. Ποια είναι τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι γίνεται με το πρόγραμμα πλαίσιο, είναι η πύλη προς την αριστεία στηρίζει αυτή την κινητικότητα του ταλέντου και τη διεθνή συνεργασία έτσι ώστε να διατηρήσουμε και να οικοδομήσουμε την αριστεία. Λοιπόν, να σας πω πως πρώτα απ' όλα σε επίπεδο συνεργατικών ε, έργων και κυρίως των πυλώνα που έχει να κάνει με τις κοινωνικές προκλήσεις, να σας πω πως ο βαθμός στον οποίο αυτές οι συνεργασίες είναι εκτός Ευρώπης είναι αρκετά χαμηλός. Δηλαδή η συνεργασία που λαμβάνει η χώρα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι συνήθως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τόσο πολύ εκτός. Οπότε, για τη συνεργασία με τα τρίτα μέρη περιορίζεται αρκετά. Γίνεται με πολλή συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό έχει βοηθήσει το πρόγραμμα πλαίσιο και δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για παραπάνω συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών μελών. Και επίσης υπάρχει το εξής θέμα. Τι θα γίνει με το Brexit. Ποιος θα συνεργάζεται με το Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα χάσει από αυτούς που συνεργάζονται σήμερα και τι περιθώριο δημιουργείται και αν θα είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με το Ηνωμένο Βασίλειο όταν θα βρίσκεται εκτός προγράμματος ε, πλαισίου. Και γι' αυτό το κοιτάξαμε ε, για να δούμε ε, τι συνέβη με το Ενωμένο Βασίλειο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και εκεί ποιε χώρε συνεργάζονται περισσότερο με το Ενωμένο Βασίλειο. Και πάλι εδώ βλέπει κανεί πω είναι οι πιο ισχυρέ χώρε. Δανία, για παράδειγμα, Νορβηγία, κάτω χώρε, Γερμανία, Σου... Ελβετία, που συνεργάζονται οι πολλοί με το Ηνωμένο Βασίλειο και αν φύγει από την εξίσωση θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε επίπεδο συνεργασία. Η Ιρλανδία επίσης και αυτό είναι ε, εδώ ένα θέμα και αυτές θα είναι οι χώρες οι οποίες θα επηρεαστούν. Δεν θα χάσει δηλαδή μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο το γεγονό ότι θα έχει λιγότερε δυνατότητε συνεργασία, αλλά και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι χώρε οι οποίε ε, πλήττονται περισσότερο και θα έχουν ε, μεγαλύτερε δυσκολίε συνεργασία, μια και θα βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο θέμα είναι το πώ είναι κανεί ελκυστικό στα ιδιαίτερα ταλέντα. Μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο ε, δίνουμε τέτοιου είδου δυνατότητε και έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο, μια και πρόκειται για επιχορήγηση που πηγαίνει σε μεμονωμένους ερευνητές για να μπορούν να μετακινηθούν και ε, αυτό επιτρέπει στο ταλέντο να κυκλοφορεί ελεύθερο στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε πως ε, στο Συμβούλιο αυτό υπάρχουν αρκετές χώρες ε, και εδώ εστιάζουμε μόνο στην αριστεία. Πολλές χώρες λοιπόν πάνε πάρα πολύ καλά και αυτό και πάλι συμπεριλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπετε όμω πω οι επιτυχίε του Ηνωμένου Βασιλείου σε μεγάλο βαθμό βασίζονται στη δυνατότητα προσέλκυσης ταλέντων. Και πάλι λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληγεί σοβαρά από το γεγονό πω δεν θα μπορεί ή τουλάχιστον πολύ πιο δύσκολο να προσελκύσει ταλέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τι χώρε που στέλνουν πολύ κόσμο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία για μια φορά ακόμα λοιπόν βλέπουμε χώρες οι οποίες σε κάθε βαθμό θα έχουν λιγότερο δυνατό, λιγότερες δυνατότητες να στείλουν επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά να τους επαναπροσλάβουν. Στο πρόγραμμα πλαίσιο ε, επιτρέπεται αυτή η δυνατότητα της προσέλκυσης ταλέντων, αλλά ε, βασικός κόμβος στο Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως το Brexit σε αυτό να μας επηρεάσει. Αυτό ήταν ε, λοιπόν ως τελευταία διαφάνεια. τώρα για τις επιπτώσεις και ποιες εγώ πιστεύω ότι θα έχει το Brexit για το Horizon Europe. Να σας πω πως και πάλι είναι σημαντικό να εστιάσουμε στην οικοδόμηση της αριστείας έτσι ώστε να είμαστε στην αιχμή του δώρατος, να εστιάσουμε λοιπόν στην αριστεία αλλά και με ανοιχτό πνεύμα, παγκοσμιοποίηση, προσέλκυση ταλέντων, συνεργασία με τους καλύτερους εταίρους, όλα αυτά είναι κομμάτια που θα γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε κάποιο βαθμό και με τις συνδεδεμένες χώρες και με τρίτα κράτη. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ρόλο τον οποίο θα παίξει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι συνδεδεμένη χώρα, θα είναι τρίτη χώρα, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να είμαστε αρκετά ανοιχτοί, έτσι ώστε να προσελκύουμε τα ταλέντα και να συνεργαζόμαστε. Με τον τρόπο αυτό θα οικοδομήσουμε την αριστεία και θα μείνουμε κι εμείς ε, πραγματικά στην κορυφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την ε, ε, ομιλήτρια που μας μίλησε για ένα ανησυχητικό πλαίσιο εξέλιξης της έρευνας. Το λόγο έχει η κυρία Μάης που θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις του Brexit στον ορίζοντα, αλλά σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας. Yes. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σε αυτή τη συνάντηση. Εγώ εκπροσωπώ την ε, Λίγα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Έρευνας. Είμαστε ένα δίκτυο 20 πανεπιστημίων σε 12 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, Πέντε μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο και 2 από την Ελβετία. Δεν ξέρω αν φαίνεται ε, στη διαφάνεια. Τα πανεπιστήμια αυτά είναι το Cambridge, η Oxford, το Imperial στο Λονδίνο, το University στο Λονδίνο, το Εδιμβούργο και η Γενέβη και η Ζηρίχη από την Ελβετία. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως είναι συνδεδεμένα ε, με το πρόγραμμα ε, πλαίσιο επειδή είναι στην Ελβετία. Η όργανωσή μα, χαράσει πολιτική ε, και ε, έρχεται εδώ στις Βρυξέλλες να μιλήσει για πολλά θέματα έρευνα, τριτοβάθμιας εκπαίδευση και καινοτομίας. Μόλις επέστρεψα από την συνάντηση των Πριτάνεων των 23 πανεπιστημίων. Ήμουνα στο Δουβλίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τα μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκεί και εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δραστήρια. Και μάλιστα πρέπει να σας πω πως έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, όπως γίνεται από το 2016 και μετά συζητάμε το Brexit είναι ε, κάτι στο θεματολόγιο μας και το συζητάνε πάντα οι Πριτάνες γιατί είναι σημαντικό για όλους μας τα μέλη από το Ηνωμένο θέλουν να παραμείνουν μέλη της ε, ΛΕΡΟΥ, του συνδέσμου μας, να συνεχίσουν να είναι κομμάτι του προγράμματος πλαισίου και για μας βέβαια είναι καλοδεχούμενοι και είναι και ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη δική μας ένωση και βεβαίω θα παραμείνουν στο δικό μας δίκτυο. Τούτου λεχθέντος αυτή τη στιγμή χτίζουν εταιρικέ σχέσεις σε όλη την Ευρώπη με όλη την υπηρετική Ευρώπη έτσι ώστε να διατηρήσουν τους συνδέσμους που έχουν και που τους είναι τόσο προσφυλείς για το μέλλον, ε, σε μια, ένα κόσμο μετά το Brexit. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μπω κατευθείαν στο θέμα. Τίποτα δεν άλλαξε από την πρώτη δήλωση που κάναμε το 16, αμέσως μετά το Brexit και το δημοψήφισμα. Στηρίζουμε ε, τα μέλη μας, στηρίζουμε τη δέσμευσή τους στην Ευρώπη και θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως το αποτέλεσμα μιας επαναδιαπραγματευόμενης ε, σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιτρέψει η συνεργασία μας να συνεχίσει, να υφίσταται για να είμαστε πάντα δραστήριοι, για να έχουμε πάντα συνεργασία με τα μέλη αυτά, ε, γιατί μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε μια επικερδή για όλους κατάσταση. Διαφορετικά, χαμένοι θα βγούμε όλοι. Δεν είναι τόσο απλό. Υποβάλαμε ε, το μήνυμα αυτό και το επαναλάβαμε και σε μια δήλωση φέτος, το Μάιο, μετά την δήλωση της κυρίας Μέη, όπου επανέλαβε την επιθυμία του Εμένου Βασιλείου να έχει πλήρη σύνδεση με το Horizon Europe μετά το Brexit. Εμείς στη Λέρου πιστεύουμε πως τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο θα λυθούν από τα πανεπιστήμια και από άλλους ακαδημαϊκούς κύκλους με συνεργατικό πνεύμα, με αποτελεσματική συνεργασία, διάσυνεροιακά, με ανοιχτή επιστήμη, ανοιχτή καινοτομία που θα εφαρμόζονται με τρόπο ανοιχτό και προβάσιμο για όλους. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο που θα επιτρέψει στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι ε, βασικός ε, εταίρος στο δικό μας οικοσύστημα των ακαδημαϊκών Ινστιτούτων στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επίσης και τα 27 κράτη-μέλη, να κάνουν ε, να θέσουν στις διαπραγματεύσεις για το Brexit την ε, καινοτομία και την έρευνα ως κορυφαία προτεραιότητα για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν σε αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία ε, στην έρευνα, ακόμα και μετά το Brexit. Αναγνωρίζουμε πως είναι δύσκολο να παραδοθεί αυτό το αποτέλεσμα, γιατί θα πρέπει να γίνει αρκετή πρόοδος σε κάποια πολλά άλλα σημεία των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Αλλά όπως είπε ε, και η προλαλή σα καθηγήτρια έχει να κάνει με την, με την κινητικότητα των ερευνητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για μας, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και μετά τον Brexit. Μετά τη δήλωση του Ιουνίου θα δείτε πως ε, τον Ιούλιο ε, εκδώσαμε 12 βασικά μηνύματα για τον Brexit και την κινητικότητα στην Ευρώπη. Καλωσορίσαμε το μήνυμα της Πρωθυπουργού Μέη και υποβάλαμε και σχέδια για το σχέδιο έκθεσης που δεν είναι πια σχέδιο των εισηγητών ε, Νίκα και Έλερ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα από τα βασικά μηνύματα ήταν πως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία και καλωσορίσαμε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το κάνει στα πλαίσια του Horizon Europe. Επίσης, θέλουμε ε, να γίνεται τη δυνατότητα να είναι κανείς συνδεδεμένο μέλος του Horizon Europe για όλα τα κράτη που έχουν γειτονική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, και να έχουν πλήρη πρόσβαση. Και θα πρέπει και η Ελβετία να έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί τις ίδιες ε, διατάξει με το παρελθόν και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνδεθεί αν κάποιες οικονομικές ε, προϋποθέσεις ε, γίνουν σεβαστές. Στα κομβικά μηνύματα του Ιουλίου θα δείτε ότι προτείναμε για κάποιες τροπολογίες έτσι ώστε να φαίνεται και αυτό στους κανόνες μας. Επίσης, Είπαμε πως Λερού δεν στηρίζει τον περιορισμό της πρόσβασης ε, σε κάποιους δικαιούχους, δηλαδή να είναι μόνο οι δράσεις Μαρή ε, Κιουρί και ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο μήνυμα που είχαμε στην αρχή του μήνα. Αυτό το είδαμε με 13 άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα ε, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το Caesar EUA, Coimbra, The Guild και άλλα πανεπιστήμια. Δηλαδή ε, ένα ευρύ φάσμα πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη. Με τις πρόσφατες ε, εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι υποβαθμίζεται ένας βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και όπως αναφέρεται και στο κείμενο, το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να συνεχίζει να ορίζει τις προδιαγραφές αριστείας στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει ότι η κυρία Γκέιγκεν Queen θα πρέπει να τονίσει ότι το Horizon Europe θα πρέπει να παραμείνει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχει σχέση με τη συνοχή της Ευρώπης. Και μια φορά ακόμα λοιπόν είμαστε κατά των προτάσεων ε, στο να περιορίσουμε την πρόσβαση σε τρίτες χώρες Και το είπαμε και σύμφωνα με τα όσα έγιναν στην Επιτροπή Ήτρε σήμερα το πρωί, γιατί αυτά όλα για μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά όταν ακούγονται. Επίσης, ένα τελικό σχόλιο θα ήθελα να κάνω για το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να παροτρύνω τα ε, κράτη-μέλη να προχωρήσουν ε, όπω και οι θεσμοί το συντομότερο δυνατόν. Και το λέω στου θεσμού γιατί έχουμε να κάνουμε με τι πολιτικέ διαπραγματεύσει για τον Brexit και υπάρχουν και άλλα δύσκολα σημεία στο ίδιο το Horizon Europe που δεν είναι σχετικά με αυτό. Αλλά θα ήταν πραγματικά αρνητικό αν το Horizon Europe ξεκινήσει καθυστερημένα Αυτό είχε γίνει και στο Horizon 2020 και δεν ήταν καθόλου ε, καλό. Μπορεί να υπάρχει κάποιο κενό σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα θέλαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, ε, έτσι ώστε ε, να ξεπεραστεί το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αν διαφυσβήτητα κάποιο κενό θα έχουμε. Ό,τι και να γίνει μετά τη Σύνοδο την Κυριακή και ό,τι και να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, είναι δεδομένο πως όλα αυτά θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επόμενες φάσεις και το είδος του Brexit ε, θα λάβουν χώρα. Και ελπίζω πως όλοι θα κατανοήσουν πως χρειαζόμαστε ε, κάτι να συμβεί γρήγορα, γιατί μια καλή, ε, καλή οριοθέτηση των θεμάτων της έρευνας ε, θα δώσει και κάποια μηνύματα θετικά για τις γενικότερες σχέσεις μας μετά το Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Η τρίτη ομιλήτρια είναι η καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Κουίπερ. Σίγουρα δεν έχω προφέρει καλά το όνομά σας που θα μιλήσει για τις επιπτώσεις του Brexit μέσα στα πλαίσια της ε, βιομηχανίας και του τομέα των φαρμακευτικών σκευασμάτων που είναι ύψης σημασίας για την υπηρετική Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και την Επιτροπή σας που μας ε, κάλεσε σήμερα το απόγευμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας δώσω την επιτυχή και την απόψη της φαρμακοβιομηχανίας, γιατί για μας από την αρχή την διαπραγματεύσεων για τον Brexit λέγαμε ότι για τις εμπορικές ε, ε, ενώσεις και τις εθνικές ενώσεις Εξ αρχή ε, ήμασταν σε επαφή με του συναδέλφου μα από τον Εμμανό Βασίλειο και με τη φαρμακοβιομηχανία για την ανάγκη να κρατήσουμε τη συνεργασία μεταξύ μα. Και νομίζω ότι για μα ω κλάδο δεν μα απασχολεί μόνο ο επιχειρηματικό κλάδο. Φυσικά πολλά ακούμε στα μέσα ενημέρωση για το κόστο για τι εταιρείε και τι βιομηχανίε ε, σε ό,τι αφορά το κόστος ε, με την κατάσταση λόγω Brexit. Για μας όμως εκπροσωπώντας ε, μια, ε, ένα κλάδο που τον απασχολεί η υγεία του κόσμου, πάντα λέγαμε ότι είμαστε ξεχωριστός κλάδος. Και το τονίσαμε αυτό εξ αρχής τον κύριο Μπαρνιέ, ότι δεν είμαστε μια ένα κανονικό κλάδο και παρακαλώ αυτά συνεχίζουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίση, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούμε ω κλάδο στην πολιτική διακήρυξη τη Κυριακή, ακριβώ επειδή είναι ο χαρακτήρα του κλάδου μα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη και στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει μεταξύ τη Ευρώπη ε, των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα και η ανάπτυξη είναι η ουσία της βιομηχανίας μας και βλέπετε τι δαπανούμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη σε σχέση και με άλλους τομείς, 35 δισεκατομμύρια και έχουμε 750.000 άτομα τα οποία απασχολούμε στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι ύψη μιλάμε και τι μεγέθη μιλάμε. Πέρα λοιπόν από την επικέντρωση στις αλυσίδες προμήθειας, όπου συνεργαζόμαστε και με πολλές ε, θεατρικές εταιρείε, γιατί προετοιμαζόμαστε και για ένα σενάριο χωρίς συμφωνία και φαντάζεστε ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές σε αφορά προμήθειες, γιατί κάθε μήνα 45 εκατομμύρια φάρμακα έρχονται από το ΕΒ Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 37 εκατομμύρια αντίστροφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Και η έρευνα όμω είναι στην ατζέντα μα, όχι μόνο οι προμήθειε. Και αυτό θα πρέπει να μείνει, να παραμείνει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά σε έναν κλάδο που έχει μεγάλη παγκόσμια διάστηση. Δεν έχει νόημα να αποσυνδέσουμε όλες τις προτάσεις που έχουν προσπαθήσει που γίνουν τα τελευταία 30-40 χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί βασικό παράγοντα και γι' αυτό θα πρέπει να παραμένει συνεργασία. Και το Ηνωμένο Βασίλειο συμβάλλει περίπου 20% στην ε, συνολική έρευνα και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο κράτος μέλος που το 2014, αν δεν κάνω λάθος, ε, ξεκίνησε ένα Υπουργείο ακριβώς για αυτές τις ε, επιστήμες ζωής. Ε. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να παραμείνει αυτή η κατεύθυνση. Και κοιτάμε λοιπόν και τις επερχόμενες ευρωεκλογέ, τι χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία του ευρώ. Είναι σημαντικό γιατί κάθε ένα ευρώ το οποίο προέρχεται από τα ταμεία επενδύσεων προσελκύει 6 ευρώ από ιδιωτικό, τον ιδιωτικό κλάδο. Αυτό σημαίνει κάτι. Ελπίζουμε λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η συμμετοχή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η ανταγωνιστικότητα του κλάδου, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο παίζει σημαντικό ρόλο. 20% λοιπόν τη έρευνα τη ανάπτυξη μεταξύ 2007 και 2016. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίση έχει μοναδικέ εγκαταστάσει έρευνα που επίσης ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Επιστήμη, γιατί πραγματικά είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Δεν ωφελείται μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελείται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από τις ε, ερευνητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το κέντρο Midline και άλλα κέντρα που διδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το Ηνωμένο Βασίλειο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην πρωτοβουλία για τα γενοτομικά φάρμακα IMI. E και εδώ βλέπουμε πόσο σημαντική πάλι είναι συνεργασία και αυτή η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ πανεπιστημίων, ακαδημαϊκού κόσμου, έρευνα και ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντική, σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το ε, ευάλωτο οικοσύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί ο σύνδεσμος αυτός και στον δρόμο και μετά το Brexit. Για το Venture Capital αναφέρατε τι ε, γίνεται και είπατε ότι αυτό σημαίνει και σημαντική απόδοση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πέρα από τον αντίκτυπο του Brexit. Προφανώς το Brexit δεν έχει μόνο αντίκτυπο στην ε, έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά και στην κινητικότητα των επιστημόνων. Γιατί και πάλι στα πλαίσια της ε, πρωτοβουλία IMI, όπου έχει γίνει μεγάλη δουλειά, μπορούμε να πούμε ότι πολλές από τις εταιρείες μας, που είναι παγκόσμιες κλίμακας εταιρείες, απασχολούν πολύ κόσμο και έξυπνο κόσμο και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την ευελιξία και μετά το Brexit σε όλο τον κόσμο. Δεν αρνούμε την πολιτική πραγματικότητα, αλλά λέω απλά ότι θα πρέπει και μετά το Brexit να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ των ε, ανθρώπων αυτών για να μην ε, προκληθούν εμπόδια για τη σταθερομία των ατόμων αυτών. Ως ε, FPA λοιπόν, ως ε, φαρμακευτική βιομηχανία υποστηρίζουμε ένα σύστημα το οποίο θα διευκολύνει την κινητικότητα και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι γρήγορο και ξεκάθαρο γιατί ας δούμε φυσικά τι θα μας φέρει αυτή η τελική συμφωνία αποχώρησης Ολοκληρώνουμε τώρα στην τελική μας ανάλυση για να δούμε ποιες θα είναι συνέπειες και στον τομέα της κινητικότητας. Αλλά κάποια από τα πρώτα παραδείγματα τα οποία ακούσαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας ήταν, έδωσαν και πολλές ελπίδες για την ταχύτητα και την αμεσότητα του συστήματος. Αν λοιπόν μια ευρωπαϊκή, αν κάποιος έχει την επιλογή να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο να μείνει στην Ευρώπη ή να έχει μια παγκόσμια θέση. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεται η απόφαση αυτή για τους επιστήμονες, για τον λόγο λοιπόν αυτό το, το τονίζω εκ νέου. Ελπίζουμε να είναι ξεκάθαρο και ρεαλιστικό το σύστημα που θα αποφασίσουμε γιατί και πάλι εξαρτώμαστε από την κινητικότητα, εξαρτώμαστε από προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης όχι μόνο για τους ερευνητέ και τους τα συμφέροντα αυτών, αλλά και τις μελλοντικέ γενιές, γιατί περίπου 60.000 φοιτητέ από ευρωπαϊκές χώρες είναι καταχωρισμένοι σε άνωτα ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και 6.500 εξ αυτών είναι σε επίπεδο μεταπτυχιακό. Καταλαβαίνετε λοιπόν και πάλι για τη μεγέθεια μιλάμε και πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί αυτό το σημαντικό οικοσύστημα και για τις επόμενες, επερχόμενες γενιές. Άρα, ασφαλώς ε, ξέρουμε ότι σε λίγες ημέρες θα έχουμε και την τελική συμφωνία αποχώρησης και την πολιτική διακήρυξη και ξέρουμε σήμερα ότι έλαβε χώρα η ψηφοφορία για τον Ρεζοντάι Ευρώπη στην Επιτροπή σας. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι και το Συμβούλιο θα πρέπει να συζητήσει τμήματα της συμφωνίας αυτής και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει υπόψη του τα στοιχεία αυτά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στον οριζόντα Ευρώπη και υπολογίζω ότι θα υπάρξει και θα επικρατήσει και κάποια κοινή λογική στο το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί δεν φτάνει μόνο η δουλειά από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή σας αλλά χρειάζεται κοινή λογική και σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου. Να μην ε, μπλοκαριστεί η συνεργασία επειδή δεν θα μπορούν ενδεχομένω να ηγούνται τη ε, έρευνα. Και εδώ πρέπει να φέρω και την πολιτική πτύχη, αλλά να κλείσω λέγοντα ότι η συμμετοχή στον Ορίζοντα Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στα πλαίσια τη ε, έρευνα και τη ανάπτυξη και τη κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική σημαντικές πτυχές για μένα το παγκόσμιο κλάδι, όχι μόνο για μας ως επιχειρήσεις και ως κλάδο, αλλά και στην τελική ανάλυση για τη δημόσια υγεία και για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για αυτή την άκρος ενδιαφέρουσα παρέμβαση και για τα συμπεράσματά σας. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον ε, συνάδελφο Νίκα γιατί μίλησε, μιλήσαμε για το Horizon Europe και ήταν βασικός εισηγητής του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Συμφωνώ με αυτά που είπατε και θα αισθανόμουν καλύτερα αν υπήρχαν αυτές οι παρουσιάσεις πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. Γιατί νομίζω ότι δεν υπήρχαν ε, όλα τα στοιχεία πριν από το δημοψήφισμα και αυτό το βλέπουμε εκ του αποτελέσματος γιατί δύο χρόνια μετά μπορούμε να αποτιμήσουμε τις ε, συνέπειες, τις αρνητικές συνέπειες του εάν, πώς, γιατί. Η αλήθεια είναι μία. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πούμε «Μα τι κάνετε». Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να μπει σε μία διαδικασία ε, τι ε, θα συνέβαινε αν είχαμε διαφορετικά δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος του Horizon Europe. Ε, αν αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να μπει στη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τι θα γίνει, ποιο καθεστώς θα το διέπει. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς, θα το αποφασίσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό ε, είναι σαν να χτυπάμε μια ανοιχτή πόρτα. Και αυτό το λέω εις εισηγητής. Ήρθα σε επαφή με την κυβέρνηση του Ενωμένου Βασιλείου, με τις οργανώσεις, ε, με, ε, ήρθα σε επαφή με το πρόγραμμα Guild Caesar και ούτω καθεξής. Μου είπαν το ίδιο. Μου είπαν ότι αυτό είναι πολύ αρνητικό και για τις δύο πλευρές. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στο Horizon Europe, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για τη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, τους ακαδημαϊκούς, τους φοιτητές, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι τίποτα στο χέρι μας. Ό,τι μπορούσαμε το αποφασίσαμε. Εμείς ψηφίσαμε να συμμετέχει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο στο Horizon Europe αν αποσυρθεί εξαρτάται από την ίδια τη χώρα. Υπάρχει και η πολιτική της ε, επιλεκτικότητας. Θα μπορέσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες, ίσως να πείσουμε τους Βρετανούς εταίρους ότι θα διαπραγματευτούμε να παραμείνουν μέρος του προγράμματος ή όχι. Άκουσα για αυτά που είπατε ως προς την ελεύθερη ε, διακίνηση των ερευνητών. Είναι βασική αξία για όλους τους πολίτες. Μιλάμε για τους ερευνητές, για τους γιατρούς και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ακολουθούμε λάθος δρόμο, αλλά δεν επιβάλλω εγώ το κανονιστικό πλαίσιο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να προσεγγίσετε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και να αρχίσετε τις διαπραγματεύσεις. Γιατί συζητήσαμε με τον Μισελ Μπαρνιέ και με τον Κίφερ Χόρφστατ και αυτά που ακούσαμε δεν ήταν ενθαρρυντικά. Δυστυχώς. Αυτό για να έχετε μια εικόνα του τι σημαίνει Brexit. Έτσι ώστε κανένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να μην έχει διαφορετική θέση και δεν είχε. Σήμερα ψηφίσαμε ομόφωνα όλες οι πολιτικές ομάδες να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Horizon Europe. Μην κοιτάτε λοιπόν το πρόγραμμα, μην κοιτάτε τι, τους άλλους όρους για τις συνδεδεμένες χώρες, για τις τρίτες χώρες, για να δείτε ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτό θα ήθελα να το καταστήσω απόλυτα σαφές. Δηλαδή ε, ε, δεν χρειάζεται να ε, ασκήσετε πίεση εδώ ως λόμπιστε. Εμείς έχουμε ανοιχτές πόρτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στο Horizon Europe γιατί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αποχωρήσει τότε το θέμα επαφίεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. σε σχέση με την αριστεία και το μέλλον. Αυτό που κάνουμε στο Horizon Europe είναι να ενισχύσουμε τα κριτήρια αριστείας, να είναι πιο ορατά, αλλά και να υπάρχει διαφάνεια, να δείξουμε γιατί επιλέγησαν αυτά τα σχέδια, γιατί χρειάζεται καλύτερη, καλύτερη πληροφόρηση όλων των φορέων. Είδαμε τα αποτελέσματα, τα δεδομένα και βλέπετε όλα τα προγράμματα τα οποία φαίνονται με διαφάνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και θα πρέπει να καλωσορίσουμε αυτή τη διαφανή προσέγγιση που έχει προβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε σαφή κριτήρια για το τι μπορεί κανείς να κάνει αν δεν είναι ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί η αριστεία αναγνωρίζεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει σημασία απλώς να αξιώνουμε την αριστεία, αλλά να δείχνουμε ότι πληρούμε τα κριτήρια της αριστείας. Δεν φασιζόμαστε πουθενά αλλού και νομίζω ότι όλοι είσαστε υπέρμαχοι αυτής της προσέγγισης. Μιλήσατε επίσης για τους δικαιούχους. Horizon Europe, ε, the money αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι τα χρήματα προέρχονται από τους Ευρωπαίους ε, φορολογούμενους και θα πρέπει να καταδείξουμε πώς ε, δαπανούμε και πώς κατανέμουμε τα χρήματα. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο πραγματικός δικαιούχος να φαίνεται σαφώς. Δηλαδή, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Δεν θέλω να δώσω τα ονόματα των χωρών αυτή τη στιγμή. Αλλά εσείς μπορείτε να τις επιλέξετε γιατί παρατάσσονται πολλές χώρες. Ένα πράγμα είναι να υπάρχουν πανεπιστήμια και ερευνητές ένα συνεργατικό πλαίσιο και άλλο να δίνει κανείς 50.000 σε, στις ΜΜΕ. Γιατί πολλοί είπαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εμείς δεν κρίνουμε ότι αυτό είναι σκόπιμο γιατί υπάρχουν, υπάρχουν οι εθνικές επιδοτήσεις. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο ε, κριτήριο που είναι η προστασία του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συμφέροντος με βάση αυτά που έχει ορίσει το ελεγκτικό συνέδριο, που ελέγχει τι συνέβη με αυτά τα χρήματα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει αν πρέπει δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο να ταξιδέψει ανά τον κόσμο για να δει πώς δαπανήθηκαν αυτά τα 50.000 ευρώ. Και αυτό είναι το θέμα που αφορά τους μεμονωμένους δικαιούχους. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ε ανά τον κόσμο από το Horizon Europe. Και ό,τι και να κάνουμε θα πρέπει να ξέρουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να ελέγξει την ε, πραγματική δαπάνη των χρημάτων. Όλα τα άλλα ζητήματα την χάνουν υποστήριξης και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, διότι με περιστοιχίζουν δύο Βρετανοί συνάδελφοι, Βρετανίδες μάλλον, εκδεξιών και εξεβονίμων. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό το τι συμβαίνει. Άκουσα τα πανεπιστήμια, την φωνή των ερευνητών και ξέρω ότι νιώθουν πολύ άσχημα. Ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ξέρουμε ποιες θα είναι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι καθαρό κέρδος, αλλά καθαρή απώλεια. Ξέρουμε το αποτέλεσμα εν μέρη, το οποίο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση. Και στις 27 χώρες. Αλλά πιστεύω δεν μπορούν να υπάρχουν σύνορα στην αναγνώριση αριστείας. Η μακροπρόθεσμη έρευνα στον τομέα του καρκίνου, η ανάπτυξη της γραφήν, του γραφήν που ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, αυτό που δεν κάνουν οι τράπεζες είναι να επενδύουν μακροπρόθεσμα, γιατί μέχρι σε 7 χρόνια θα πρέπει να έχουν κεφαλαιοποίηση και αυτό που καταφέρνουν ε, ορίζοντας ε, Ευρώπη και τα λοιπά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρόγραμμα είναι ακριβώς να κάνουν μακροπρόθεσμη επένδυση. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους επιστήμονες να κινούνται ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη για να ε, κατακτήσουμε εκ νέου την κορυφαία θέση για την Ευρώπη σε παγκόσμιο προσκήνιο, να εργαστούμε με τα καλύτερα ταλέντα μας, να συνεργαστούμε και να πω ότι ο Ντάν ήταν αυτός που επέμενε στον ορίζοντα Ευρώπη προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι απόλυτο μέλος, ισότιμο μέλος και το ψηφίσαμε σήμερα το πρωί με υποστήριξη από όλα τα κόμματα, όλες τις πολιτικές ομάδες. Επίσης, συμφωνώ ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε και να στραφούμε στον κόσμο στις τελευταίες φάσεις της συμφωνίας. Θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι τους είπαν ψέματα. Αν σας πω ότι ήθελα να πάω σε μεγάλο σταθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μιλήσω για τέτοια θέματα αλληλεξάρτησης ε, μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα ενέργειας. Και τι έκανε λοιπόν ο σταθμός αυτός πριν από το δημοψήφισμα. Ήταν τόσο υπεύθυνοι που ανταυτού εξέπεψαν την ε, άρνηση της αλλαγής του κλίματος του UKIP. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να απευθύνω. Συγγνώμη μετά από μια μεγάλη εισαγωγή είναι σε τι βαθμό πιστεύετε ότι σας ακούν, σας εισακούν από πλευρά τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τερέζα είναι στις Βρυξέλλες για διαπραγματεύσει την ώρα που μιλάμε, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε όλα τα άτομα στην επικρατεία τη να υποφέρουν λόγω του Brexit. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ λοιπόν σήμερα. Άλλο ε, Μία άλλη Yeah. Uh, so another... Άλλος ένας συνάδελφος από τη Βρετανία, λοιπόν, που υποστήριξε το να παραμείνουμε, θα λάβει το λόγο. Λοιπόν, Τέλος πάντων, θα ακολουθήσω και εγώ τα όσα είπε η Τερέζα και είναι πολύ παρόμοια η δική μου οπτική. Να σας πω πως αυτή τη στιγμή ε, θέλω να επανέλθω στο σημείο για τα πακέτα με τα 45 και τα 37 εκατομμύρια. Άκουσα από φαρμακευτική εταιρεία την περασμένη εβδομάδα πως Όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της Αριάννα Γκράντε, δεν υπήρχαν αρκετοί επίδεσμοι και γάζες στο Μάντσεστερ για τους 500 τραυματίες. Πολλά από τα άτομα αυτά ήταν παιδιά και έφεραν με αεροπλάνο επιδέσμους και γάζες και γι' αυτό κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και ήταν όλα αυτά τα υλικά, τα φαρμακευτικά μέσα σε λίγες ώρες. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς δεν ρώτησε τίποτα, ούτε στα αεροδρόμια, ούτε οπουδήποτε και δεν χρειάστηκε να περάσουμε από καμία διαδικασία έτσι ώστε να γίνει ό,τι χρειάζεται για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που με ε, εντυπωσίασε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ντάν γιατί με έχει ανεχθεί που τον ενοχλώ συνέχεια γιατί θέλω το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι όσο δυνατόν πιο, πιο βαθιά μέσα στο Horizon Europe και να έχουμε μια μελλοντική σχέση στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Αλλά ο Ντάν έχει απόλυτο δίκιο. Δεν το δημιουργεί το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι οι ευρωπαϊκές οντότητες, είναι οι Βρετανοί. Με τις κόκκινες γραμμές και με όλα αυτά. Ελπίζω πραγματικά πως το αποτέλεσμα του της εβδομάδας και με το μελλοντικό ε, πλαίσιο που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την έρευνα με την λεπτομερή συμμετοχή στο Horizon Europe να τα καταφέρουμε. Όμως θα πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, αναφερθήκατε την περίπτωση όπου δεν θα έχουμε συμφωνία, το no deal. Νομίζω αυτό είναι το μόνο για το οποίο υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στην ε, Βουλή ε, είναι ότι είναι αντίθετη με τη μη συμφωνία. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, αν τελικά φτάσουμε εκεί, δεν θα μας επιτρέψει ε, να αυτοτραυματιστούμε σε αυτό το βαθμό, γιατί αυτό βέβαια θα έχει και κάποιες παρεπόμενες θα επιφέρει και παρεπόμενες ε, βλάβες. Νομίζω πω τελικά οι ενήλικοι θα τα καταφέρουν και θα κυριαρχήσουν και κάποιο είδους λογική θα μπει στη συζήτηση. Οπότε προτείνω σε όλους να μην χρησιμοποιούμε την ε, μη λύση, τη μη συμφωνία ως όπλο εκβιασμού για την κινητικότητα είναι πολύ ζωτική σημασία. Και πάλι έχει δίκιο Ντάνι. Η ελευθερία κίνησης είναι μια γενική αρχή. Και είναι μια αρχή η οποία δεν είναι και τόσο λίγο δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν γίνεται μια άμεση έρευνα για την ελευθερία μετακίνησης και κυκλοφορία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθω η μέτρηση είναι θετική αρκετά πάνω από το 50%. άλλαξε μετά το δημοψήφισμα, αλλά δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα και πριν. Και μπορώ να βρω πάρα πολλού λόγου να σα εξηγήσω, αλλά πρέπει να σα πω πω υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο και αυτό έχει να κάνει πάλι με το τι θα κάνει η Βρετανική κυβέρνηση για τα όσα έχουν υποθεί ε, μέχρι τώρα με την απόλυτη πάυση της ελεύθερης κυκλοφορίας και δεύτερον για το πώς λειτουργεί η μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και το μισθολογικό. Γιατί αν κοιτάξουμε αυτόν τον κλάδο, γιατί μιλάμε για του διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που μετακινούνται, το πρόβλημα το πρώτο να έχεις φοιτητέ που να συμπεριλαμβάνονται στους αριθμούς των μεταναστών και δεύτερον να έχεις αυτά τα μισθολογικά θέματα που λαμβάνονται υπόψη είναι εξαιρετικά προβληματικό για τούτο το τον κλάδο. Συμφωνώ 100% με ε, τον ΝΙΚΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την μακροπρόθεσμη ε, χρηματοδότηση και την πρόθεση σε αυτήν. Θα κλείσω λέγοντας πως ε, για τις ε, ε, επιστήμες. Ε, συμφωνώ με τα όσα είπατε. Έχω συνεργαστεί με πολλές από αυτές τις ενώσεις των θετικών επιστημών και νομίζω ότι είναι υπέρ όλων μας, όπως συμβαίνει και με τις σπάνιες ασθένειες κτλ. Οπότε για να επαναλάβω και εγώ τα όσα είπαν οι δύο προλαλήσαντες, η πραγματικότητα της κατάστασης σήμερα είναι πολύ πιο σαφής. Δεν πιστεύω πως το πακέτο ή η συμφωνία απόσυρσης είναι επαρκής πρόταση για τη χώρα μου. Δεν θεωρώ πως η μη συμφωνία είναι λύση την οποία θα προκρίνουμε. Άρα λοιπόν αρχίσουν και χάνονται οι εναλλακτικέ λύσεις, το μόνο δίκαιο και το λέω αυτό γιατί ήμουν συνδικαλίστρια. Εγώ ποτέ δεν θα συμφωνούσα μια τελική συμφωνία χωρίς να ζητήσω από τα μέλη μου αν συμφωνούν. Και νομίζω ότι είναι δίκαιο τελικά να επιστρέψει κανείς στο λαό και να του πει «Ωραία, Μα σας είπαμε αυτό, τα πράγματα άλλαξαν, αυτή είναι η πρόταση. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα έχουμε μπροστά μας. Είναι δίκαιο και σωστό εσείς που ψηφίζετε να έχετε την ευκαιρία τώρα που έχετε ενημερωθεί να κάνετε τις επιλογές σας. Και γνωρίζω πως όταν κάναμε το πρώτο δημοψήφισμα ε, στις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια όλοι ψήφισαν να παραμείνουν. Γιατί τα πανεπιστήμια κατάφεραν να μιλήσουν με τις κοινότητες τους και κατάφεραν να εξηγήσουν ποια είναι η πραγματικότητα που είναι στο τραπέζι. Πιστεύω το να συνεχίσουμε με όλο, πιο περισσότερη, όλο μεγαλύτερη ενημέρωση, αυτή ακριβώς η περισσότερη ενημέρωση θα μας οδηγήσει στο να κάνουμε μια επιλογή ε, ενημερωμένη που θα πηχεί τα καλύτερα συμφέροντα ε, για το μέλλον της χώρας μου. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις, ήταν άκρος ενδιαφέρουσες και νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, θέλει, θα θελήσει να συνεργαστεί μαζί σας. Ε, ακούσαμε πολλά που αποτελούν προβολές στο μέλλον, ότι πω, πω μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί εκείνο, όλα αυτά τα έχουμε ακούσει. Όταν δούλευα στο Westminster, όταν, το μεγάλο, όταν η Μεγάλη Βρετανία δεν μπήκε στην Ευρωζώνη, μας είπαν ότι τότε θα πληγούμε ιδιαίτερα, μας περίμενε ζωφερό μέλλον. Δεν μπήκαμε στην Ευρωζώνη και ευημερίσαμε οικονομικά και είμαστε η πέμπτη η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Μας είπαν ότι μετά το δημοψήφισμα θα χάνονταν πολλές θέσεις εργασίας, θα είχαμε καταστάσεις επίγουσας ανάγκης από δημοσιονομικής πλευράς. Δεν ε, συνέβη κάτι τέτοιο, διότι αυτοί που ήθελαν να παραμείνουν ε, έκαναν, προέβησαν μάλλον σε αυτή την κινδυνολογία. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, μας είπαν, αλλά όλα αυτά ήταν κινδυνολογία. Διαψεύστηκαν. Μιλήσαμε για την επιμελητία. Ε, εγώ ασχολήθηκα στον τομέα της επιμελητίας και της μεταφορών μέσα στα πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού της βιομηχανίας. Ξέρω πως δουλεύει η αλυσίδα εφοδιασμού και μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο προβληματικά όπως τα παρουσιάζεται. Η Μεγάλη Βρετανία έχει εμπόριο με πολλές ε, χώρες μέσα τα πλαίσια του ΠΟΕ. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Θα το ξεπεράσουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρξει συμφωνία, σε περίπτωση no deal, τα πράγματα θα έχουν καλή έκβαση. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα να τα δούμε με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Υπάρχει πολύ καλό μέλλον για το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον κόσμο. Άλλοι βουλευτές είπαν πω πω φεύγετε και ούτω κάθε εξής. Εμένα πολλοί ευρωβουλευτές μου είπαν πω, πω μακάρι να φεύγαμε μαζί σας, μακάρι να αποχωρούσαμε και εμείς. Άρα τα πράγματα είναι αμφίδρομα. Εγώ προσβλέπω στο μέλλον μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάν για δεύτερο δημοψήφισμα γιατί έχασαν στο πρώτο. Ήταν το μεγαλύτερο δημοκρατικό δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα βρίσκονται σε μια κατάσταση άρνησης. Η Βρετανική κυβέρνηση είπε θα εφαρμόσουμε το αποτέλεσμα. Δεν θα διενεργηθεί άλλο δημοψήφισμα και άλλο και άλλο μέχρι να έχουμε το αποδεκτό αποτέλεσμα. Εάν σταματήσετε το αποτέλεσμα με ένα νέο δημοψήφισμα, αυτό θα είναι επονίδιστο. Αλλά το είδαμε να γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν θα συμβεί όμως στη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ προσβλέπω σε ένα λαμπρό μέλλον. Συνάδελφοι, θα ήθελα να μην θίγεται το θέμα Brexit ως προς τις επιλογές. Να παραμείνουμε στο θέμα μας. Γενική ε, έκκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι καινούριο εδώ και έχω μια ερώτηση να κάνω. Καταρχά, μου προκάλεσε έκπληξη. Είμαι στο νόσο, είμαι λίγο στερετικό. Είμαι ο μόνο εδώ που ε, υπερασπίζομαι τη μεγάλη χώρα της Μεγάλης Βρετανίας. Είμαι ο δεύτερος μόνο. Ο προηγούμενος ε, ομιλητή είπε αυτά που σκεφτόμουν. Γιατί αυτό που με απασχολεί είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω. Όλοι το λένε, το είπαν και οι δύο κυρίες προηγουμένως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να μείνει. Αναρωτιέμαι λοιπόν και διαρωτώ μα, μα πώς τι άλλο έγινε. Και τώρα έχουμε το Brexit ε, πρωτοθυρών. Ξέρω ποια είναι η απάντηση η στάνταρ απάντηση. Αυτός ο διάολος, ο Νάιτζελ Φάρατζε, κατάφερε να ξεγελάσει το μεγάλο έθνος. Αν είναι τόσο διαβολικός, σατανικός πια, τι να κάνουμε. Μου προκάλεσε έκπληξη όμως κάτι άλλο. Πραγματική έκπληξη μου προκάλεσε το γεγονός ότι το Brexit είναι μόνο του. Γιατί πολλές άλλες χώρες έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν λέω κατά πόσον το δέχομαι ή όχι. European Union. I think about Ιταλία και άλλες χώρες να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μήπως θα πρέπει να ρεμίσουμε και να δεδοτηθούμε. κατά πόσον εμείς, η Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο, τι κάναμε και προέκυψε αυτό, τι κάναμε λάθος, πού σφάλαμε. αυτό το εσωτερικό δρόμο που πήραμε. Όλα αυτά δεν θα μας βοηθήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Αν ε, έρθει η στιγμή που πούμε ότι κάτι κάναμε λάθος και αν εμείς ήδη παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθη, Ίσως ε, τότε να ελπίσω ότι κάποια μέρα θα σταματήσουμε να κάνουμε λάθη και θα ζούμε σε μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κατανοούμε αλλήλους και ούτω καθεξής. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αυτή τη στιγμή να ασκήσουμε κριτική. Ίσως να μην έχουμε επαφή με τον κόσμο έξω στους δρόμους όπως θα έπρεπε. Μήπως είμαστε υπερβολικά ελιδιστές. Ίσως να αντιλαμβανόμαστε μόνο διαρρετικά τέτοια project και όχι τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Αλλά ο κόσμος εκεί έξω τι θέλει. Θέσεις απασχόλησης, να μην φοβάται, καλή εκπαίδευση. Το ακούσαμε σήμερα το θέμα της καλής εκπαίδευσης και με συγχωρείτε. Πού το είδατε αυτό την τελευταία φορά. Και στον εμένα βασίλειο. Το θέμα της εκπαίδευσης ε, δεν υπάρχει πλέον πουθενά. Αν δεν ε, ασκήσουμε ειλικρινή αυτοκριτική, αν δεν διορτηθούμε, μα πού κάναμε λάθος, γιατί εμείς φταίμε, το Brexit θα επαναληφθεί. Σε Συγχαρητήρια σου, Βρετανούς, όπως και να έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ασκήσουμε και λίγη αυτοκριτική. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Σας ευχαριστώ για όλες τις υποδείξεις. Εγώ δεν ε, θα ήθελα να γίνει το Brexit, γιατί ξέρετε ότι προέρχομαι από την ε, Ιταλία. Εγώ άκουσα ε, συζητήσεις με πάθος, ζωηρές συζητήσεις και συζητήσεις που σχετίζονται με την καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων. Μιλάμε για υγεία. Πέρα από την έρευνα και την ε, καινοτομία, όταν μιλάμε για την υγεία, μιλάμε για τις ε, καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Νομίζω λοιπόν ότι ο λόγος μας ήταν συνεκτικός και οι συνομιλήτριές μας ίσως ε, θα θέλαν να αντιδράσουν εντάχει, γιατί έχουμε και πολλά άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη που θα μας απασχολήσουν. Και σε ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους ομιλητές που μίλησαν από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ως προς το Brexit για την έρευνα έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι για να αποδώσει η επιστήμη θα πρέπει να προτάξουμε την αριστεία που θα πρέπει να είναι ανοιχτή στα ταλέντα και τη συνεργασία. Γι' αυτό το Brexit αποτελεί ε, οριστική απώλεια. Τώρα θεωρώ ότι δεν μπορείτε να συγκρίνετε το θέμα με τη γενικότερη έρευνα. Θα υπήρχε απόλυτο κέρδος αν παρέμενε το Ηνωμένο Βασίλειο στον ερευνητικό τομέα. Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο και δεν προέκυπτε το Brexit, αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση. Κατανοώ όμως ότι υπάρχουν ε, ε, πολιτικές επιτακτικές ανάγκες, γι' αυτό θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τη ζημία. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε εξαιρετικούς ε, ερευνητές και επιστήμονες, κάτι το οποίο σημαίνει ανοιχτά σύνορα. Το ίδιο αφορά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τους εκπροσώπους. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η αριστεία. Η ανοιχτή συνδρομή της αριστείας. Μην ξεχνάμε αυτή την κατάσταση win-win, δηλαδή απόλυτου κέρδους εκεί όπου μπορούμε. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων, που είναι απαράβατος όρος για να έχουμε μία κατάσταση ολικού κέρδους. Και τέλος, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην κοιτάμε μόνο το το χρηματοοικονομικό σκέλος, πόσα θα πάρουν οι μεν και οι δε. Το ζήτημα είναι ποιο είναι το ολικό ευεργέτημα από την επιστήμη. επιστήμη. Εκεί θα πρέπει να εστιάζεται η συζήτηση για να έχουμε το, το βέλτιστο στο δυνατό ευεργέτημα. Τέλος. Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις μετά το Brexit, κατά πόσο θα είναι μια συνδεδεμένη τρίτη χώρα, το, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει την πλαισίωση γενικότερα με όλες τις χώρες, δηλαδή πόσο ανοιχτοί είμαστε στις άλλες χώρες ε, γενικότερα. Ωραία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι. Η επόμενη ομιλήτρια. Thank Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη όμως. Για διάφορου λόγους. Να αναφέρω αυτό το θέμα των μονοδικαιούχων. Για μας ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό προγράμματα όπως ε, οι δράσει ε, Marie και των Ευρωπαίων, τα ευρωπαϊκά προγράμματα να συνεχίσουν να υπάρχουν και παρά το γεγονός ότι το ERC και πολλές από τις δράσεις του MSCA δίδονται ως επιχορήγηση σε ένα άτομο, η έρευνα στις πιο πολλές περιπτώσεις σήμερα δεν γίνεται από ένα άτομο μόνο του. Σχεδόν πάντα αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια. Αν λοιπόν εξετάσετε μια α, επιχορήγηση επιδότηση ERC, δεν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο είναι σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια χώρα μόνο. Συνήθως περιτραγυρίζεται από μια διεθνή ομάδα ερευνητών μεταδιδακτορικών. Να το έχετε λοιπόν αυτόν υπόψη σας όταν μιλάμε για μόνο δικαιούχου. Και άλλο ένα σύντομο σημείο θα ήθελα να επισημάνω. Είμαι επικεφαλής των δράσεων τη Συμβουλευτική Ομάδα για τα Υποτροφίε Μαρία για τον ορίζοντα τη Ευρώπη. Και συζητάμε, αν και φυσικά δεν εμπίπτει στον τομέα αρμοδιότητά μα, ε, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε σκέψει για το πώ ε, το ορίζοντα Ευρώπη θα μπορούσε να καλύψει και τη Μαρία Φυσικά η Μαρία αποτελεί ένα πρόγραμμα αριστείας και αυτό θα πρέπει να παραμείνει ως στοιχείο. Αλλά υπάρχει σωστή προσοχή προκειμένου να συνεχιστούν οι δράσεις επέκτασης στα πλαίσια του προγράμματος Μαρικυρή. Η Ευρώπη θα είναι πιο δυνατή αν ο κόσμος έχει δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε όλη την Ευρώπη. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι αμοιβαίως επωφελέ αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει στα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ. Και τελευταία εισηγήτρια να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή και νομίζω και ελπίζω να ξεκαθάρισα ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι υπέρ μια συμφωνία για μελλοντική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη των 27 χρειάζονται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Και το σημαντικό στοιχείο θα ήθελα να επαναλάβω προς τους Βρετανούς Ευρωβουλευτές ότι είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρώπη των 27 κατανοούν τα στοιχεία αυτά, αλλά μαζί με τις βρετανικές οργανώσεις είμαστε σε επαφή και με την νέα βρετανική κυβέρνηση και πραγματικά από την αρχή του σταθήξαμε τα θέματα αυτά. Προφανώς το Brexit είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Πέρα λοιπόν από τα θέματα αυτά πίσω από τα προσκήνιο, υπάρχει μεγάλη κατανόηση, αλλά ενδεχομένω να μην υπάρχει κατανόηση όταν τα βλέπετε τα πράγματα αυτή κανεί απ' έξω. Έχετε δίκιο φυσικά ότι εμά, ε, ως ε, κλάδος η αλυσίδα προμήθεια δεν αποτελεί θέμα γιατί είμαστε παγκόσμια, παγκόσμιος κλάδος. Ωστόσο, έχουμε, αποτελούμαστε από επιχειρήσεις και στα δύο χρόνια που έχουμε δεν αρκούν για να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα μεταφερθούν ε, Ένα γενικότερο θέμα είναι ότι στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για σύγκληση ακόμα και συμπεριλαμβανομένη του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία 30-40 χρόνια. Τώρα λοιπόν, όταν θα καταστεί τρίτη χώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να κινηθούμε προς την ε, πλευρά της απόκλησης. Αυτό είναι διαφορετικό. Και από την παγκόσμια προπτική νομίζω ότι ξεκαθάρισα ότι για όλους μας είναι πιο θετική η σύγκληση και όχι η απόκληση. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα καταρχήν να μας ε, δώσετε τις διαφάνειες και να παρουσιάσετε, να κάνετε μία ανακεφαλαίωση της παρουσίασης θα βοηθούσε τους συναδέλφους γιατί έχουν σημασία όχι μόνο οι διαφάνειες αλλά και η συλλογιστική σας. Να μας στείλετε μία συγκεφαλαίωση με ε, το βασικό σας σκεπτικό, τη συλλογιστικής σας. Ως προς τον οργανισμό ε, Marie Curie θα ήθελα εφόσον συνεργάζεστε με την Επιτροπή να μας πείτε πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτό το πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια της αριστείας για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μία πιο ενισχυμένη συνέργεια. Γιατί ε, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μία συστημική προσέγγιση. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα ήταν άκρος ενδιαφέρον και αν έχουμε και το γραπτό σας υπόμνημα θα το διανύμουμε. Λοιπόν, όσο αποχωρούν ε, οι καλεσμένες μας, έχουμε ορισμένες ε, εκθέσεις του Καρίνς που δεν βρίσκεται εδώ. Ας δούμε λοιπόν με ε, την ετοιμότητα από αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Φλάβιο θα μας μιλήσει για το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ θα είμαι πολύ σύντομος. Μετά τον ε, δεύτερο τριμέρι και ορισμένα τεχνικά σημεία είχαμε πολύ καλή έκβαση των διαπραγματεύσεων και θα είναι καλύτερη αύριο, κατά τον, κατά τον τρίτο τριμέρι. Επίσης, ε, ως πως το ΆΣΕΡ θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να επιμείνουμε για τον ορισμό μεθοδολογίας που θα τεθεί σε συζήτηση. Η σχέση Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων. Αυτό αφορά τα κέντρα περιφερειακού συντονισμού και μέσα στα πλαίσια του μοντέλου για την αναδιάρθρωση εθνικών σχεδίων για να υπάρχει συγκρισιμότητα, καθώς και ε, συναθρηστικά στοιχεία για τον συντονισμό και τις αντισταθμίσεις μέσα στα πλαίσια της ε, αλληλεγγύης για την αντιστάθμιση και αποζημιώσεις. Ε, νομίζω ότι θα φτάσουμε σε θετική έκβαση, αλλά δεν υπάρχει υπάρχει ολοκλήρωση των ε, θεμάτων που αφορούν όλες τις πτυχές της ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε το Regional Coordination Center και την ε, ομοιογένεια και συντονισμό εθνικών και περιφερειακών σχεδίων. Αυτά τα προγράμματα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και άτυπων διαπραγματεύσεων για τον αυριανό τριμερή. Δεν έχουμε φτάσει σε τελική συμφωνία με το Συμβούλιο, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία και ευχαριστώ τους τι διότι με υποστήριξαν ουσιαστικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Μπούζεκ που ήταν παρόν. Σας ευχαριστούμε. Εάν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, θεωρούμε ότι έχει κλείσει αυτό το θέμα. Ε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τζανονάτο και ο κύριος Πέτερσεν θα μας μιλήσει για τον τριμερή σε σχέση με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί ο τρίτος τριμερής διάλογος θα γίνει απόψε, θα ξεκινήσουμε στις 8. Οι δύο έχουν ήδη γίνει και δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κλείσουμε το θέμα απόψε δυστυχώς γιατί θα χρειαστούμε σχεδόν σίγουρα ακόμα μία συνάντηση που μάλλον θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον απόψε προσπαθούμε να κλείσουμε κάποια από τα άρθρα που είναι ακόμα ανοιχτά. Επίσης, θα ευθυγραμμιστούμε με τα αποτελέσματα των ε, διαπραγματεύσεων που γίνονται για την ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εκεί τρέχουν διαπραγματεύσει για τη σχετική οδηγία και δεν έχουν ακόμα κλείσει. Οπότε προοδεύουμε μεν, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ό,τι είχαμε αρχικά προβλέψει, όμως περιμένουμε προσδοκία τον τριμερή διάλογο απόψε. Ελπίζω ότι και εκεί κάπως θα προχωρήσουμε. Καλή επιτυχία για απόψε. Έχουμε ένα τελευταίο σημείο Πρόκειται ε, για την ενημέρωση της αποστολής Ήτρες στο Μιλάνο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 18 εντάχει ε, επισκεφθήκαμε την ΕΞΠΟ για να δούμε τι έγινε στη μεγάλη αυτή έκθεση και εμβαθύναμε τα προγράμματα που αφορά, συγγνώμη, ε, αφορούν ένα μεγάλο κέντρο, ένα μεγάλο πόλο νοσοκομείων και κέντρα ε, βιομηχανικού, βιομηχανικής ανάπτυξης, ένα τέτοιο πόλο. Μιλήσαμε για την ψηφιοποίηση του βιομηχανικού τομέα επισκεφθήκαμε την Ίσπρα, ε, το κοινό κέντρο ερευνών και είδαμε ότι υπάρχει δυνατότητα εμβάθυνσης των ε, αποφάσεων και της εφαρμογής τους και τέλος έγινε μία επίσκεψη στην έδρα ε, Λεωνάρντο σε αυτή τη μονάδα που έχει μεγάλη σημασία για την τεχνολογική ανάπτυξη της Ιταλίας. Στην περιφέρεια της Λομβαρδίας μιλήσαμε για το ε, κέντρο, το κοινό κέντρο ερευνών και είδαμε, επισκεφτήκαμε το, ένα innovation hub δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν που θα μπορούσε να μας μιλήσει για αυτό τον κόμβο καινοτομία στη Λομβαρδία που βοηθά τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και παράλληλα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας αυτόν τον κόμβο καινοτομίας. Κάτι το οποίο είναι άκρος ενδιαφέρον. Αφορά την ενεργειακή απόδοση, το τομέα της υγείας και ούτω καθεξής. Ε, πρόκειται για 200 startups. Έτσι είχε λοιπόν η επίσκεψή μας οι συνάδελφοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Είχαμε ε, μία ε, έντονη δραστηριότητα από το πρωί ε, έως το βράδυ σε αυτή τη διημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο στις 9 για να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη και είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε μία κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Μεταφορών. Ε, στο 3 σε 50. Αλλά το ξέρετε αυτό, έτσι κι αλλιώς δεν έχουν μείνει και πολλοί για να κοινοποιώ τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο το πρωί.